Um, ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ σα αρχίσουμε. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Στην απογευματινή μας συνεδρίαση θα μιλήσουμε για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και το ΣΕΣΑΡ, την ε, τον επιχειρησιακό αντίκτυπο στις αποστολές ε, της ΚΕΠΑ και τις ε, στρατιωτικές ικανότητες. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μαουρίτσιο Καστελέτη που είναι Δηματάρχης για τον Ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, Γενικό, Γενική Διεύθυνση της Κινητικότητας των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Καστελέτη αντικαθιστά τον κύριο Μπάλντουιν που ζητά συγγνώμη ε, για την απουσία του γιατί βρίσκεται στην Ελλοδαπή. Ε, δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Λουκ Τικέτ, ο Διευθυντής ε, για τον Ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό στη Eurocontrol. Έχουμε και τον κύριο Κάρλο Μποργκίνη, που είναι υποδιευθυντής, εκτελεστικός υποδιευθυντής ε, στην κοινή επιχείρηση ΣΕΣΑΡ και τον κύριο Τζαμπάλο Λίλο που είναι διευθυντής εξοπλισμού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Αυτοί είναι οι τέσσερις καλεσμένοι μας. Βλέπετε ότι έχουμε πολλούς Ιταλούς στο πάνελ, θα έλεγα η <laughs> και στην αίθουσα. Ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ε, είναι ένα θέμα που το έχουμε ήδη συζητήσει στην υποεπιτροπή μας και τον Οκτώβριο, από ό,τι μάλλον γνωρίζετε, υιοθετήσαμε και την έκθεση για την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και μάλιστα υποβάλαμε και την δική μας γνωμοδότηση με εισηγητή τον κύριο Κυρίλοφ, ε, ε, σοσιαλιστή από τη Βουλγαρία. Τονίζει την ανάγκη συνεργασίας πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου και την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να μας κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Τους θέρμα παρακαλώ να μην ξεπεράσουν το δεκάλεπτο στην πρώτη τους παρουσίαση. Μετά θα έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις και θα μπορέσετε στα πλαίσια των απαντήσεων να αναπτύξετε τα διάφορα σημεία. Κύριε Καστελέτη, έχετε το λόγο πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά σας ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του Διευθυντή μου, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση αυτή. Θα επικεντρωθώ κυρίως στο πολιτικό πλαίσιο καθώς επίσης και στην φάση εγκατάστασης και εφαρμογής του ΣΕΖΑΡ. Αν ξεκινήσουμε από τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το ΣΕΖΑΡ αποτελεί ένα τμήμα της πολιτικής της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Πρόκειται για τον τεχνολογικό πυλώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να εκμορδενήσει τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και κυκλοφορίας και αν δείτε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό θα καταλάβετε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους θέλουμε να εμπλέξουμε το στρατιωτικό τομέα. Πρώτον, στα πλαίσια της προμήθειας των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποιες στρατιωτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα στην Ιταλία οι μετρολογικές υπηρεσίες παρέχονται από την πολεμική αεροπορία ή κάποια αεροδρόμια παρέχουν αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, στρατιωτικά αεροδρόμια παρέχουν αεροναυτιλιακές υπηρεσίες στον πολιτικό τομέα, μη στρατιωτικό τομέα. Επίσης ο στρατιωτικός τομέας με τη σειρά του χρησιμοποιεί υπηρεσίες της πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή ακολουθεί τους κανόνες της GAT, της Γενικής Ενέργειας Κυκλοφορίας. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της χρησιμοποίησης ε, ενός κοινού πόρου, δηλαδή του ενάηρου χώρου. Και το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί προκύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Προφανώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χώρο για εμπορικέ πτήσεις, αλλά πρέπει και η πολεμική αεροπορία να μπορεί να χρησιμοποιεί τον ενέργειο χώρο για τις ανάγκες ασφάλειας και άμυνας. Στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και στα πλαίσια του ΣΕΖΑΡ έχουμε κάποιες απλές πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τον τίτλο της σημερινή μας συζήτηση βλέπουμε ότι θα μιλήσουμε για την επίπτωση του ΣΕΖΑΡ του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού στις και τις στρατικές ικανότητες της ΚΕΠΑ. Το ΣΕΣ και το ΣΕΖΑΡ είναι καταρχάς ε, πολιτικές μη στρατικές πρωτοβουλίες και λογικά δεν έχουν αντίκτυπο στο στρατικό τομέα. Πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες ε, εκπονήθηκαν στα πλαίσια της διαχείρισης του ε, ενέργειου χώρου από μη στρατικές πτήσεις. Επί της αρχής λοιπόν το ΣΕΖΑΡ δεν θα πρέπει να έχει άμεσες επιπτώσεις στις στρατικές ικανότητες και ούτε θα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αεροπορία εκπονεί τις αποστολές της. Είδαμε όμως ότι υπάρχει μια κάποια έμεση επίπτωση γιατί όπως σας είπα και πριν από λίγο ο στρατιωτικός τομέας μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στον πολιτικό και το αντίστροφο. Και είπαμε ότι ο στρατιωτικός τομέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΓΚΑΤ, τη γενική ενέργεια κυκλοφορία και οι δύο κλάδοι χρησιμοποιούν ένα κοινό πόρο τον κοινό ενέργειο χώρο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εμπλέξουμε τον στρατιωτικό κλάδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου στα πλαίσια της πολιτικής ΣΕΖΑΡ. Αυτό αποτελεί μια προστιθέμενη αξία της πολιτικής που ακολουθούμε, να καταφέρουμε να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη στρατιωτική, στρατιωτική κοινότητα στην όλη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και για το ΣΕΖΑΡ. Αυτό ήδη συμβαίνει μέσω διαφόρων επιτροπών που ήδη συνεδριάζουν και φέρνουν τους δύο κλάδους μαζί και θα αναφερθεί στο ζήτημα αυτό και ο κύριος Μποργκίνη κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του και θα ακούσετε επίσης και την άποψη του Eurocontrol που είναι άλλωστε ένας οργανισμός που φέρνει μαζί και το στρατιωτικό και τον πολιτικό κλάδο. Όσον αφορά τώρα το ΣΕΖΑΡ και την εφαρμογή του, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στον κανονισμό αυτό ο εγκρίθηκε το Μάιο του 2013 κανονισμό 409 του 2013. Ξέρετε ότι το ΣΕΖΑΡ έχει τρει διαφορετικέ φάσει. Τη φάση του καθορισμού, τη φάση τη ανάπτυξη και τη φάση τη ε, εφαρμογή. Η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο, δημιούργησε το ATM Master Plan. Ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η φάση της ανάπτυξης από την ε, κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ, ενώ η φάση της εγκατάστασης εφαρμογής θα ξεκινήσει λογικά του χρόνου. Αν μελετήσετε τον κανονισμό αυτό θα δείτε ότι έχει συνταχθεί δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο που μπορεί να δραματίσει ο στρατιωτικός τομέας. Υπάρχει διαιτελογική σκέψη παριθμών 19 η οποία αναφέρει ότι το ΣΕΖΑΡ θα πρέπει να συντονιστεί με την στρατιωτική πλευρά και ότι το ΣΕΖΑΡ δεν θα πρέπει να έχει αρνητική επίπτωση στις στρατιωτικές επιπτώσεις. Τι εννοούμε με αυτό. Θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, ενδεχόμενες αυτές επιπτώσεις γιατί ενδεχομένως το ΣΕΖΑΡ να θέσει κάποιες απαιτήσει για την πολιτική χρήση, τη μη στρατιωτική χρήση, που μπορεί στη συνέχεια να έχουν κάποιες επιπτώσεις στο στρατιωτικό κλάδο και αναφέρομαι σε χρηματοοικονομικές κυρίως επιπτώσεις. Επίσης υπάρχει ένας ορισμός για, τον, ε, για τους ε, stakeholders, του στρατιωτικούς, στο άρθρο 2 σημείο 9 αναφερόμαστε σε φορείς παροχής υπηρεσιών και χρήστες τόσο από τον πολιτικό όσο και από τον στρατιωτικό τομέα. Επίσης, στο πρώτο τμήμα του καονισμού προσπαθούμε ακριβώς να δούμε τι πρέπει να εφαρμόσουμε και αναφερόμαστε στα common projects, στα κοινά σχέδια. Ποιος θα πρέπει να εφαρμόσει τα σχέδια αυτά και πότε και πού ακριβώς θα πρέπει να εφαρμοστούν στην ε, διαδικασία αυτή του καθορισμού της τεχνικής πτυχής ε, της νέας αυτής αντίληψης που θα πρέπει να εφαρμοστεί, λέμε ότι ο στρατικός κλάδος θα πρέπει να εμπλακεί και αυτός πλήρως και γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά στην, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ε, εντοπιστεί ως βασικός ε, συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου μέσω αυτού του οργανισμού να καταφέρνουμε να μαθαίνουμε τις απόψεις του στρατικού κλάδου. Έπειτα τίθεται και το ζήτημα της διακυβέρνησης που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα. Έχουμε το επίπεδο της πολιτικής, το επίπεδο της διαχείρισης και το επίπεδο της εφαρμογής. Στο επίπεδο της πολιτικής, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μία ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προωθήσει τη συμμετοχή των στρατιωτικών της στρατιωτικής κοινότητας όσο το δυνατόν περισσότερο και στο άρθρο αυτό που αναφερόμαστε στο πολιτικό επίπεδο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας λέγεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα διευκολύνει το συντονισμό των απόψεων που προέρχονται από τον στρατικό κλάδο και θα υποστηρίξει τις απόψεις τις αμυντικές των κρατών μελών καθώς επίσης και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς στρατιωτικές οργανώσεις και κρυμμένα στο ΝΑΤΟ. Και θα μπορούμε στη συνέχεια τις, εφαρ... τις απόψεις αυτές να τις υλοποιήσουμε στα πλαίσια της φάσης εγκατάστασης του ΣΕΖΑΡ. Βλέπετε λοιπόν ότι προβλέπεται μέσω συγκεκριμένων διατάξεων η έμπρακτη συμμετοχή του στρατιωτικού κλάδου στο ΣΕΖΑΡ. Προφανώς πρέπει να υπάρχει όμως μια καλή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να τροφοδοτήσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε για να εμπλακεί ο στρατιωτικός κλάδος. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ακόμα ένα τμήμα του κανονισμού το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο με τη στρατιωτική πλευρά και να φέρουμε πρώτα στην συμμετοχή της στρατιωτικής πλευράς σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο της διαχείρισης και στο επίπεδο της εφαρμογής. Όσον αφορά την διαχείριση, τη διακυβέρνηση, θα υπάρχει ένας επικεφαλής. Δεν είναι ακόμα γνωστό ποιος θα αναλάβει την ε, διαχείριση του, του επίπεδου αυτού. Πάντως θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαρθρωθεί στο επίπεδο αυτό να δυνατόν καλύτερα συνεργασία με τον στρατιωτικό τομέα. Δηλαδή η ε, διαδικασία της εφαρμογής εγκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει στον το περισσότερο και το στρατικό κλάδο. Στη συνέχεια προσπαθούμε να δούμε πόσο η στρατιωτική κοινότητα μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στο επίπεδο του συντονισμού μέσω των ε, deployment managers, των διαχειριστών της φάσης εγκατάστασης. Μία άλλη πρόκληση έχει να κάνει με τον καθορισμό των προτύπων που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτή τη φάση της εγκατάστασης, της εφαρμογής. Και γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε στρατιωτικά πρότυπα. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τον υφιστάμενο στρατιωτικό εξοπλισμό και να δούμε στη συνέχεια αν μπορεί να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στα στρατιωτικά πρότυπα και τα μη στρατιωτικά πολιτικά πρότυπα. Να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δύο συστήματα μπορούν να συνεργαστούν χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, εξασφαλίζοντας μια πλήρη διαλειτουργικότητα. Τέλος, το επόμενο στάδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε είναι η διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων αυτών που θα αποτελέσουν ε, τμήμα της φάσης εγκατάστασης. Προβλέπεται ένα συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο θα προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του οποίου θα προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιε τεχνολογίε μπορούμε να εφαρμόσουμε, αρχή γενομένες από του χρόνου. Υπάρχει ήδη ένα ενδεικτικό κατάλογο των τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν και κάποιε από αυτέ τι τεχνολογίε μπορούν ενδεχομένω να επηρεάσουν το στρατιωτικό κλάδο. Είναι σημαντικό το λοιπόν για μας να καταλάβουμε με απόλυτη σαφήνεια πώς οι τεχνολογίες αυτές μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν το στρατιωτικό κλάδο, τη στρατιωτική κοινότητα και σε ποιο βαθμό. Και από χρηματική πλευρά συγκεκριμένα, δηλαδή ποια θα είναι η χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί από τον στρατικό κλάδο και πώς μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο ο στρατικός κλάδος να υποστηρίξει και αυτός από τη δική του την πλευρά την φάση της εγκατάστασης. Θα υπάρχει πάλι και εδώ απόλυτο συντονισμό, γι' αυτό χρειαζόμαστε την εμπλοκή και των δύο πλευρών, πολιτικού και στρατιωτικού, και είπα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υφιστάμενη τεχνολογία. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι τήρησα το χρόνο των 10 λεπτών και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για τη Eurocontrol ε, η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή τη δημόσια ακρόαση και στο δεκάλεπτο που μου δίνετε θα ήθελα να σας αναφέρω και είναι τα επιτεύγματα ε, στη συνεργασία πολιτικού στρατιωτικού τομέα. Η προσπάθεια εναρμόνισης συνεργασίας ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Eurocontrol ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1960 για να δημιουργήσει μια πλατφόρμα μεταξύ των δύο πεδίων για να γίνει καλύτερη διαχείριση του εναέριου χώρου ε, και να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουμε τέτοια εμπειρία δηλαδή από το 1960. Και εμείς στην Ευρώπη Έχουμε πολιτικοστρατητική οργάνωση, έχουμε και τις δύο δηλαδή στη Eurocontrol, γι' αυτό και μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις απαιτήσεις και των δύο χρηστών σε μια ενιαία προσέγγιση. Μάλιστα, οι νέε αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα διαχείριση ενέργεια κυκλοφορία πρόσθεσαν την ιδέα ενός δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου που κρίθηκε ως απαραίτητο για να επιταχυνθεί η συζήτηση και ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών της πολιτικής και της στρατιωτικής. Και με βάση αυτές τις νέες αρμοδιότητες ε, έχουμε προκλήσεις ε, και για τη στρατιωτική κοινότητα αλλά και για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. Γιατί κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υιοθετεί κανονισμούς για τη διαχείριση ενέργειας κυκλοφορίας ε, προσπαθούμε να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και πώς θα μπορέσουν αυτές να συνεχιστούν στον εθνικό εναέριο χώρο αλλά και στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, τηρώντας φυσικά ταυτόχρονα και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μάλιστα μερικές φορές οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί και για τους ε, στρατιωτικούς ε, χρήστες. Οπότε έχουμε νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας ε, για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στην εφαρμογή των κανόνων και ταυτόχρονα έχουμε την έννοια της ελαστικής χρήσης του αέριου χώρου. Αυτό δεν είναι επινόηση της Ευρώπης, έχει σχεδιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι κάτι που το έχουμε κάνει απομονωμένα. Η διαφορά είναι ότι σε εμά είναι υποχρεωτικό. Οπότε θα πρέπει από τη στιγμή που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη να αντανακλάται και στη διοργάνωση του εναέριου χώρου. Επίσης, η Eurocontrol ε, διαχειρίζεται και τα δίκτυα. Έχει και τέτοια λειτουργία η Eurocontrol. Αυτή η λειτουργία της διαχείρισης δικτύων έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίνει λύσεις και στους πολιτικούς και στους στρατιωτικούς χρήστες και μιλούμε για γενική εναέρια κυκλοφορία κυρίως. Και αυτό το εργαλείο θα θεωρηθεί και ως ε, μοντέλο για το πώς θα μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε ενιαίες λύσεις και να συντονίσουμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη διαχείριση του ενέργειου χώρου. Ένα άλλο ε, στοιχείο από το δεύτερη πρόταση για τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό είναι τα FABs, τα λειτουργικά μπλοκ ενέργειου χώρου, η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που έχουν τη νομική δυνατότητα να οργανωθούν και σε περιφερειακό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τα όρια αυτής της ε, επιχείρησης αν δεν διευκολύνουμε την διασυνοριακή συνεργασία ακόμη και σε επίπεδο FAB. Ε, κάτι άλλο που επίσης ε, αναφέρεται και δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες είναι το θέμα του Mission Trajectory, αυτή η πορεία της ε, αποστολής, η τροχιά της αποστολής. Και εδώ θέλουμε συντονισμό από επιχειρησιακή άποψη, αλλά επίσης να εκπληρώσουμε τα εθνικά κριτήρια άμυνας σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό ενός ασφαλούς σενάριου χώρου και αυτή η έννοια της ε, πορείας της αποστολής έχει σχεδιαστεί για τους στρατιωτικούς και στηρίζεται σε ένα ελαστικό ενέργειο χώρο, ένα ελαστική χρήση του ενέργειου χώρου. Θέλουμε να προωθήσουμε μία ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των αεροσκαφών. Αν έχουμε κλειστέ ζώνε άσκηση ή αν, έχουμε, αν ανοίγουν από τη στιγμή που τελειώνει μια άσκηση, θα πρέπει αυτέ οι πληροφορίε να είναι άμεσα διαθέσιμε για όλους τους χρήστες, όχι μόνο τους ε, στρατιωτικούς που θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τη ζώνη της άσκησης, αλλά και για τις ε, αεροπορικές εταιρείες που θα έχουν πια πρόσβαση σε αυτή τη ζώνη που έχει ανοίξει. Οπότε η προωθημένη ε, ελαστικότητα του ενέργειου χώρου είναι κάτι που θα εφαρμοστεί γρήγορα. Κάτι άλλο που κάνουμε στην Eurocontrol είναι να καταρτίζουμε εναρμονισμένους κανόνες για τα στρατιωτικά αεροσκάφη γιατί έχουμε εθνικές ε, διατάξεις και τώρα υπάρχει μια, μια παράκληση για ευρωπαϊκές διαδικασίες ε, διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας, ένα ελέγχου της ενέργειας κυκλοφορίας. Γιατί ε, σε προαιρετική βάση οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της Eurocontrol. Ένα άλλο θέμα είναι η δημιουργία μιας τεχνικής ε, αρχιτεκτονικής που θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ραδάρ και επίσης την ανάγκη κλεισίματος του ενέργειου χώρου για ανεφοδιασμό. Έχουμε τα μη επανδρομένα συστήματα ε, αεροσκαφών που επίσης μπορούν να δίνουν πληροφορίες ε, για τις επιχειρήσεις και αυτές μπορούν να, να ε, ανταλλάσσονται μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής κοινότητας. Γι' αυτό η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών. Επίσης σημαντική είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών εδάφους και του αεροσκάφους. Με κατάλληλη συνεργασία των δύο προγραμμάτων εγκατάστασης, ε, του πολιτικού και του στρατιωτικού, θα διευκολύνουμε και τη στρατιωτική κοινότητα. Και αυτά είναι από τα πλεονεκτήματα για τη στρατιωτική χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Η Eurocontrol αποφάσισε να εγγενιάσει ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην αρχή μιας κεντρικής υπηρεσίας και μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα είναι προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει στον ενέργειο χώρο, που υπάρχουν ζώνες άσκησης, πότε κλείνουν, πότε ανοίγουν και ούτω ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η επαναχρησιμοποίηση των στρατιωτικών ικανοτήτων προκειμένου να φτάσουμε στο κατάλληλο επίπεδο ε, επιδόσεων, ε, επιτήρησης ε, και πλοήγησης. Έτσι μπορούν οι δύο κοινότητες να εξετάσουν τις ικανότητές τους και τα στοιχεία που έχουν, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, σε επίπεδο ΦΑΠ και νομίζω ότι έτσι γίνονται καλύτερες οικονομίες. Αυτό που ε, συστήνουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας είναι στην κοινή επιχείρηση να έχουμε κοινή διαδικασία πιστοποίησης και τυποποίησης. Δηλαδή να εγκρίνεται και να χρησιμοποιείται και από το πολιτικό και το στρατιωτικό κλάδο. Αυτή η, πρόθεση που ε, αυτή η πρωτοβουλία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ελαστική και εστιάζεται στις ανάγκες των χρηστών. Οπότε, τι είναι τελικά ο, Ευρωπαίος ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ουρανός, ευκαιρία ή κίνδυνος για το στρατιωτικό κλάδο. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά αν δεν θέλουμε να χάσουμε χρήστες από το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει και πάλι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι χρήστε του χώρου και προκειμένου ο στρατιωτικός κλάδος θα συνεχίσει ελεύθερα να πραγματοποιεί τις αποστολές του και να μην περιορίζεται από κανόνες που επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες και μπορούν να έχουν παρενέργειες σε στρατιωτικούς χρήστες του ενέργειου χώρου. Και το θέμα της ε, εταιρική σχέσης ε, πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου θα ωφελήσει και τους στρατιωτικούς ε, με δείκτες επίδοσης, οικονομία καυσίμων, άμεση, άμεσο και σύντομος ε, αεροδιάγραμμος. Επίσης αυτοί οι δείκτες επίδοση μπορούν να εκπονηθούν από κοινού από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ενδιαφερομένους και να υπάγονται από αναθεώρηση και από τους δύο. Οπότε θα έχουμε όχι μόνο περιορισμούς αλλά και πολύ θετικά στοιχεία που θα μειώνουν το κόστος και την αποτελεσματικότητα των αποστολών και των πτήσεων και του στρατιωτικού κλάδου. Με τον ενίο ουρανό έχουμε την ευκαιρία και για διασυνοριακές ασκήσεις ή διασυνοριακές αποστολές. Μια πραγματική περιφερειακή συνεργασία δηλαδή, που θα είναι υποφελής και για το στρατιωτικό κλάδο. Επίσης, επαναχρησιμοποίηση των υπαρχουσών υποδομών θα ευνοήσει τη στρατιωτική κοινότητα να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες των ραντάρ ή άλλα στοιχεία ε, οι υπάρχοι υπηρεσιών πλοήγησης ε, μπορούν να δίνουν πληροφορίες ε, και στους ε, στρατιωτικούς για εντοπισμό αεροσκαφών για παράδειγμα. Βλέπετε υπάρχουν περιορισμοί αλλά υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες που θα ωφελήσουν και το στρατητικό κλάδο. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. θα ακολουθήσει ο κύριος Κάρλο Μπορκίνη. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ε, ε, ε Ακούσαμε τον Μαωρίτσιο Καστελέτη την προσέγγιση πολιτικής της συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών χρήσεων του εναέριου χώρου. Ακούσαμε για την ανάπτυξη, ακούσαμε για την εφαρμογή από την σκοπιά της Eurocontrol ε, από τα χείλη του Λουκ. Να σας εξηγήσω τώρα ε, την, την οπτική γωνιά του Σέσαρ και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ λαμβάνει χώρα μέσω από μια εταιρική σχέση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ. Σε αυτή βασίζεται. Από την αρχή προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι στρατητικοί κοιμοί θα μπορούν να συμμετέχουν στα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό προφανώς περιλαμβάνει όλη την στρατιωτική κοινότητα. Στην αρχή η εμπλοκή της στρατιωτικής κοινότητας στο πρόγραμμα αυτό γινόταν μέσω της συμβολής του Ευρωκοντρόλ που συμμετέχει προφανώς στο πρόγραμμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά σιγά όμως ο στρατιωτικός κλάδος άρχισε να συμμετέχει περισσότερο απευθείας μέσω των κρατών μελών. Έχουμε 98 στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες από 10 ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στα σχέδια ΣΕΖΑΡ και από το 2011 και μετά προσπαθούμε να έχουμε μια διευθέτηση συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ο οποίος αποτελεί κεντρικό σημείο επαφής, προκειμένου τα κράτη-μέλη και οι στρατικές οργανώσεις να μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στο ΣΕΖΑΡ και τελικά να εξασφαλίσετε κατά αυτόν τον τρόπο συμμετοχή των στρατικών αρχών σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Και αυτό ουσιαστικά υπερβαίνει τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο να εμπλέξουμε το ΝΑΤΟ και άλλους βασικούς Στρατιωτικού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά το Πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά το πρόγραμμα. Προσπαθούμε να προετοιμάσουμε αυτό το που ονομάζουμε Release 4, την τέταρτη δηλαδή φάση του προγράμματο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είμαστε σε θέση τώρα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματο Cesar και ιδίω όσον αφορά το στάδιο 1 και στάδιο 2 μπορούμε πλέον να περάσουμε σε συγκεκριμένες εφαρμογές όσον αφορά την διαχείριση ενέργειας κυκλοφορίας και θα μας σε θέση, όπως είπε και ο Προαλής στο μέλλον, να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα όσον αφορά τις πορείες, τροχές, στρατιωτικής αποστολής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε επίσης να προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί καλύτερα τον χώρο και θα είναι και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Η στρατιωτική κοινότητα συμμετέχει λοιπόν στο πρόγραμμα αυτό από την αρχή από τότε δηλαδή που πρωτοαναπτύξαμε το πρόγραμμα μέχρι τα τελευταία στάδια, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα αποτελέσματα του πρόγραμμα ΣΕΖΕΡ να μπορούν να εφαρμοστούν από το στρατοτικό και τον πολιτικό κλάδο. Θα πρέπει επίση να είναι φιλικό προ το χρήστη το πρόγραμμα, είτε είναι από το στρατοτικό ή μη κλάδο, και θα πρέπει να συνεπάρχουν και να λειτουργούν τόσο οι στρατιωτικέ πτήσει όσο και οι μη στρατιωτικέ πτήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε όχι τα αποτελέσματα μόνο της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά καταφέρνουμε επίσης να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να έχουμε μία γενικότερη διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση του πολιτικού και στρατικού κλάδου και να βρούμε κάποιες συγκεκριμένε λύσεις προκειμένου να εντάξουμε περισσότερο το στρατικό κλάδο στο πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Ο κύριο Στίρκατ πριν από λίγο αναφέρθηκε στι βασικέ αρχέ που υπογραμμίζουν το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε την τροχιά στρατιωτικής αποστολής, την ευέλικτη χρήση του νέριου χώρου. Σήμερα δεν έχουμε ευέλικτη χρήση ακόμα του νέριου χώρου, αλλά βλέπουμε ότι ε, στο μέλλον δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις όλο και περισσότερες στρατιωτικές και μη πτήσεις με τον άκαμπτο ενέργειο χώρο που έχουμε σήμερα. Επίση, προσπαθούμε να αρμονίσουμε του κανόνε ελέγχου ενέργεια κυκλοφορία. Όπω είπε και ο Μαουρίτσιο πριν από λίγο, υπάρχουν χώρε που έχουν κάποιου διαφορετικού κανόνε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια ζητήματα διάρθρωσης αρτεκτονικής. Και προσπαθούμε επίσης να, χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες αεροπορίας που, έχουμε, που διαθέτουμε σήμερα. Θέλουμε επίση να πετύχουμε ένα υψηλό επίπεδο αυτοματοποίηση, πράγμα το οποίο θα μα βοηθήσει να πετύχουμε μια καλύτερη διαχείριση τη ενέργεια κυκλοφορία και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε το προσωπικό μας να επικεντρωθεί σε κάποιες λειτουργίες υψηλότερη προστιθέμενης αξίας και να μην ασχολείται δηλαδή τόσο πολύ με το ATM, τη διαχείριση τη ενέργεια κυκλοφορίας. Το Eurocontrol αποτελεί ιδρυτικό μέλος του ΣΕΖΑΡ, το είπε αυτό και ο κύριο Στίτκατ, και θεωρούμε και εμείς ότι το ΣΕΖΑΡ αποτελεί μια ευκαιρία προκειμένου να καταφέρει ο στρατικός κλάδος να συμμετάσχει με τον καλύτερο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες πτυχές ε, που αφορούν περισσότερο το στρατικό κλάδο. Πόσο θα στοιχήσει η συμμετοχή του στρατικού κλάδου για το, στο ΣΕΖΑΡ. Υπάρχει ήδη ένα πρώτο σχέδιο όπου προσπαθούμε στο πλαίσιο αυτού στο πλαίσιο αυτό να γεφυρώσουμε τις ενέργειες έρευνας και καινοτομίας με την φάση εγκατάστασης. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τη φάση εγκατάστασης με την έρευνα και την ανάπτυξη, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και σε κάθε φορά να έχουμε, κάθε φορά να έχουμε και μια μελέτη κόστους-οφέλους ε, προκειμένου να δούμε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό και το πιο οικονομικά αποδοτικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δείτε το Master Plan του 2010, θα δείτε ότι η μελέτη κόστους ωφέλους για το στρατικό κλάδο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι ανησυχίες του στρατικού κλάδου και τη συμμετοχή του στο ΣΕΖΑΡ. Έχουμε κάποιες προκαταρκτικές πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε ακόμα μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα κρεμία ακόμα ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει ακόμα να γίνει, πεκρεμή για το μέλλον. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάντως τα ζητήματα του στρατιωτικού κλάδου ξεχωριστά. Σίγουρα θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ποιος θα είναι ο προπολογισμός, ποια θα είναι η χρηματοοικονομική συνεισφορά του στρατιωτικού κλάδου. Θα πρέπει επίσης να δούμε αν υπάρχει κάποιο επίπεδο κινδύνου, αν κάποιο επίπεδο κινδύνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να δούμε επίσης αν υπάρχουν κάποια στοιχεία του ΣΕΖΑΡ που θα μπορούσαν να διατηρηθούν αν τελικά καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πεδίο δραστηριοποίησης τόσο του πολιτικού όσο και του στρατιωτικού τομέα. Πρέπει λοιπόν να δούμε την γενικότερη οικονομική επίπτωση που θα έχει το ΣΕΖΑΡ σε περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ΦΑΜΠΗ, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από όλα αυτά, σήμερα στο πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ βλέπουμε ότι υπάρχουν επιμέρους σχέδια που έχουν να κάνουν με τη διαλειτουργικότητα πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Υπάρχουν κάποιες ad hoc μελέτες οι οποίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ και αναφέρονται στις δυνατότητες διαλειτουργικότητας προκειμένου να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τους ε, ε, υπεύθυνου για ανάληψη ε, στρατιωτικής δράση, ιδίω επικεφαλή πολεμική αεροπορία, αποφάσει που πρέπει να λάβουν. Επίση, συνεργαζόμαστε με τον Τζαν Πάολο, ο οποίος είναι υπεύθυνο εκ μέρου του EDA και συνεργαζόμαστε επίσης και στα πλαίσια του Στρατιωτικού Συμβουλίου ATM. Υπάρχει μια εμπλοκή επίσης και του ΝΑΤΟ σε διάφορα επίπεδα και προσπαθούμε να εμπλέξουμε μέσω του EDA και άλλους σημαντικούς στρατιωτικούς εταίρους. Όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν την άποψή τους σε αυτή τη διάρθρωση συνεργασίας που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και κοινή επιχείρηση ΣΕΖΑΡ. Ολοκληρώνοντα, πρέπει να σα πω ότι δεσμεύεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ να ανταποκριθεί όλο και περισσότερο στι ανησυχίε τόσο του πολιτικού όσο και του στρατιωτικού κλάδου. Αναφερόμαστε σε επιμέρου προγράμματά μα σε διάφορε πτυχέ τη συνεργασία που έχουν να κάνουν με τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, με τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρε πλαίσιο προκειμένου να μπορούν εκεί οι δύο κλάδοι, στρατιωτικό και μη, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου το ΣΕΖΑΡ να γίνεται απόλυτα κατανοητό σε όλες τις πτυχές του και θέλουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό το ευρωπαϊκό ATM Master Plan λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Ευχαριστώ. Okay, one more time. Ευχαριστώ και εγώ. Ο τελευταίος θα είναι ο κ. Τζαν Παύλο Λίλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ κοντά σας σήμερα και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το τι κάνουμε για τον στρατιωτικό κλάδο, για την υποστήριξη των αναγκών του στρατιωτικού κλάδου στο ΣΕΖΑΡ. Πριν να μπω σε λεπτομέρειες, να επεκταθώ λίγο πρώτα στην επιχειρησιακή στην, ε, σε επιπτώσει την επιχειρησιακή ικανότητα, όπως εξήγησε ο κ. Καστελέτη, και λίγο, λίγα περισσότερα από αυτά που είπε, που έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζει κανείς πώς ε, και με ποιο τρόπο επηρεάζεται ο στρατιωτικό κλάδος. Απλή ερώτηση, αλλά καμιά φορά οι απλές ερωτήσεις απαντώνται με περίπλοκα παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν μία μελέτη και για να την κάνουμε ξεκινήσαμε ομαδοποιώντας όλες τις στρατιωτικές αποστολές που μπορεί να αναλάβει ο στρατιωτικός κλάδος σε τέσσερις-πέντε βασικές ομάδες που σχετίζονται και με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΣΕΣΑΡ. Πρώτα, με προτεραιότητα δηλαδή, αναζήτηση και διάσωση ή αποστολές Scramble. Open National Air Traffic δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο. Σύνολο κανόνων δηλαδή που επιτρέπει στο στρατιωτικό κλάδο να διαθέτει προτεραιότητα στην εκτέλεση επιχειρήσεων. Αυτοί οι κανόνες είναι εθνικού χαρακτήρα. Και λαμβάνονται υπόψη από το κόνσεπτ λειτουργίας του Σέσαρ. Άρα εξασφαλίζεται εδώ η προτεραιότητα του στρατιωτικού κλάδου. Χρειάζεται βέβαια κάποια εναρμόνιση, όπως λέχθηκε προηγουμένως, των κανόνων αυτών, που όπως είπα παραμένουν υπό εθνική αρμοδιότητα. Δεύτερη ομάδα στρατιωτικών αποστολών είναι εκεί όπου χρειάζεται αποκλεισμό τμήματων του ενέργειου χώρου, όπως για παράδειγμα για ανατροφοδότηση αεροσκαφών, ανεφοδιασμό αεροσκαφών. Αυτό είναι σημαντικό βέβαια να κατανοήσει κανείς ότι δεν πρέπει να θυγεί αυτό από την εφαρμογή του ΣΕΣΑΡ. Όμως για να αξιολογηθούν αυτές οι περιοχές ο στρατικός κλάδος πρέπει να έχει τη βεβαιότητα θα μπορεί να χρησιμοποιεί το στοιχείο αυτό. Και επειδή κάνουν και εκπαίδευση σχετικά είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι η μείωση της ικανότητας εκπαίδευσης θα έχει σημαντική επίπτωση στις επιχειρησιακές ικανότητες. Τρίτη ομάδα αποστολών είναι τέτοιες που δεν απαιτούν αποκλεισμό τμήματων του ενέργειου χώρα. Για παράδειγμα, αποστολές μεταφορών που γίνονται υπό τους συνήθεις κανόνες της ενέργειας κυκλοφορίας και είναι και πιο συνήθιση. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αποστολές αυτές, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός κλάδος, όλες τις ε, υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιωθούν από την εφαρμογή του ΣΕΣΑΡ. Επίσης έχουμε δύο ακόμα ομάδες αποστολών. Πρώτον, χαμηλού ύψους πτήση και άλλες δραστηριότητες όπως βολή πυροβολικού ή ερπάς. Και εδώ χρειάζονται κάποιες ε, τοπικές προβλέψεις, αλλά πάντως είναι, επηρεάζονται λιγότερο. Ήθελα λοιπόν να επανεξετάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Ο λόγος για την εμπλοκή του στρατιωτικού κλάδου στις δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σημαντικός. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι πτυχές αφορούν όλους τους ε, στρατιωτικούς ε, φορείς. Διότι βεβαίως ο στρατιωτικός κλάδος προσφέρει και υπηρεσίες, ATM κλπ. Επίσης, οι operator των στρατιωτικών αεροδρομίων. Γι' αυτό το λόγο, χάρη στη διαθεσιμότητα και στην ικανότητα μακροπρόθεσμου οράματος των συναδέλφων μας, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν έτσι στην αρχή τα πράγματα καθόλου. Πριν από λίγα χρόνια ακόμη, ήταν αποσυνδεδεμένα τα, αποσυνδεδεμένες οι δραστηριότητες. Δεν, καμία, υπήρχε καμία γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της στρατιωτικής ε, κοινότητας. Σήμερα λειτουργούν ε, πάνω από 2.000 ε, καταδιοκτικά αεροσκάφη, 1.600 ε, ελικόπτερα, και 400 μεταγωγικά αεροσκάφη. Και αυτά βέβαια ανέρχονται στο 2% της συνολικής κυκλοφορίας, αλλά πάντως είναι μεγάλο ποσοστό. Όπως είπα υπάρχουν και ιδιαίτερες απαιτήσει, αλλά είναι βεβαίως στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας. Από την άλλη μεριά, με την Κομισιόν αναπτύσσουμε μια πολιτική όπως είπα, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος από την πλευρά της Κομισιόν, άλλωστε σας το κατέδειξαν τα λόγια των αρμοδίων της, κατανοούν πολύ καλύτερα τις ανάγκες του στρατιωτικού κλάδου και έχουμε καλύτερη συνεργασία και έχουμε εκφράσει κατ' επανάληψη την επιθυμία να συμμετάσχει ο στρατιωτικός κλάδος. Άλλωστε έχουμε προσκληθεί πάντοτε να συμμετέχουμε στα διάφορα φόρουμ και σε διάφορε άλλε μορφέ συνεργασία Υπάρχει πράγματι καλύτερη κατανόηση για τι ιδιαιτερότητε του θεωρητικού κλάδου, κυρίω για την προπαρασκευή και ανάπτυξη και πριν από την ανάπτυξη και να βρεθούν τρόποι για να υποστηριχθεί ο στρατιωτικός τομέα και χρηματοδοτικά. Αυτό και ρητά και είναι πολύ σημαντικό για μα, διότι ο Κάρλο τα εξέγησε αυτά. Από την πλευρά τώρα του στρατιωτικού κλάδου, γιατί και από τη στρατιωτική κοινότητα δεν ήταν αρχικά σαφείς οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίε. Έχουμε λοιπόν με αυτή τη συνεργασία επιτύχει καλύτερη κατανόηση του ΣΕΣΑΡ και των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρει και που εξήγησε ο ΛΥΚ. Υπάρχουν και ευκαιρίες, διότι μπορούμε να έχουμε τη, δυνατότητα βελτιστοποίησης των πτήσεων, μείωσης ε, ε, των καυσίμων, να είμαστε ταχύτερα στον ε, σκοπό μας και λιγότερο καταρκευματισμό των ουρανών. Και βέβαια πιο εύκαμπτη χρήση των, του εναέριου χώρου. Είμαστε καλύτερα συνδεδεμένοι με το ΣΕΣΑΡ και μπορούμε από ε, πρώιμη φάση ε, να παρεμβαίνουμε. Ε, είναι οι πόρτες ανοιχτές. Συμμετέχουμε και στο πολιτικό επίπεδο όπως εξηγήθηκε ήδη στην επεξεργασία κοινών project και μάλιστα στην αρχή με πιλωτικά κοινά project έχουμε συνδεθεί εκεί και σε σχέδια τα οποία τώρα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε φτιάξει ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και έχουμε και το Cesar Military Forum, το SMIF, που είναι ένα παράδειγμα συμβολής όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Η συνεργασία είναι βέβαια με όλους τους τομείς και με την Ευρωκοντρόλ και με όλους τους ε, φορείς και με την Ευρωκοντρόλ. Τώρα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Κομισιόν και για την διαχείριση, governance, σημαντικό για μας. Ο νέος κανονισμός που θα εκδοθεί, που θα ιδρύει δηλαδή τους κανόνες για το Deployment Manager Selection. Για να εκπληρώσουμε το ρόλο αυτό, αυτό που κάναμε ήταν να πείσουμε τις χώρες μέλη να ξεκινήσουν ένα ε, project κατηγορίας Α στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Δηλαδή ένα πρόγραμμα όπου συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη και μας στηρίζουν και εμάς με πρόσθετους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για να μας επιτρέψουν να παίξουμε τον ρόλο αυτό. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αρχίσουν να εργάζονται μαζί μας από την 1η Ιανουαρίου θα μεταφέρουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη του ΣΕΖΑΡ στην έρευνα και την έρευνα τεχνολογίας ώστε να μειωθεί το κόστος να διευκολυνθεί η πρόσβαση επίσης στα ευρωπαϊκά ταμεία όπως εξήγησε ο Κάρλο προηγουμένως πόσο σημαντικό είναι αυτό ακόμα και αν οι δημοσιονομικές πτυχές για το στρατικό τομέα δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί πάντως υπάρχουν κάποιες, κάποιοι χονδρικοί υπολογισμοί βασισμένοι βέβαια σε πολλές υποθέσεις δεν είναι ακριβείς, είναι και λίγο δύσκολο να παρουσιαστούν. Αλλά θεωρήστε ότι είναι περίπου τάξος μεγέθους. 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί. Άρα πολλά λεφτά. Και εκεί χρειαζόμαστε υποστήριξη. Βεβαίω, πρέπει να διευκολύνουμε και τον συντονισμό της εφαρμογής του προγράμματος, καθώς επίσης και τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκεί παίζουμε ένα ρόλο να έχουμε συντονισμό μεταξύ του προσωπικού μας και ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, πρέπει να διασφαλίσουμε, να λάβουμε υπόψη δηλαδή, ότι έχουμε ήδη ταπανίσει πολλά χρήματα για να αναπτύξουμε ένα σύστημα συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και δεν μπορούμε να δεχτούμε τώρα να απολεστούν τα χρήματα αυτά και να μην υπάρχει συμβατότητα με το σύστημα. Γι' αυτό και θα ενισχύσουμε, θα, θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Τώρα, το ΣΕΣΑΡ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει να άρουμε το θέμα αυτό στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με βασικό μήνυμα να διασφαλιστεί ότι η αμυντική κοινότητα και οι ιδιαιτερότητές της θα ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα ε, ενιαίου ευρωπαϊκού ορανού και όχι μόνο στη τεχνολογική πτυχή του. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Σιγά σιγά έχουν προσέλθει και άλλα μέλη της ε, Υποεπιτροπής. Θα ακούσουμε ερωτήσεις, είμαι βέβαιος. Όλοι αναφερθήκατε και στο χρηματοδοτικό. Και εμείς ως Κοινοβούλιο βέβαια είμαστε εν μέρη τουλάχιστον ε, υπεύθυνοι για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και μάλιστα έχουμε και δικαίωμα συναπόφασης θα σας ρωτήσω λοιπόν για τα χρήματα. Μας είπαν ότι οι αρχικές προβλέψεις είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στρατιωτική πλευρά του συνολικού κόστους περίπου 13 δις. Είναι αλήθεια τα ποσά αυτά. Υπάρχει περίπτωση να κατέβει καθόλου το ποσό αυτό και πώς εάν ναι. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Ο Γκάλερ τώρα, συντονιστή του Λαϊκού Κόμματος. Προσοχή, προσοχή, Γερμανός, λέει στα Ιταλικά ο κύριο Γκάλερ. Ακριβώς εδώ θέλω να έλθω και εγώ, γιατί είναι το κρίσιμο σημείο. Διακόπτει ο, ο κύριος Γκάλερ αναμένοντα να φορέσω τα ακουστικά. Αυτό λοιπόν έλεγα είναι το κρίσιμο σημείο. Ακούστηκε μια τάξη μεγέθους από τον κύριο Λίζεκ των 4 δισεκατομμυρίων. οι εθνικές αεροπορίες πολεμικές δηλαδή στρατιωτικές είναι διατεθειμένες να πετάξουν με τη βάση αυτή που έχουν γίνει ενδεχομένως ήδη μέχρι τώρα επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή όταν μας λέτε ότι υπάρχει πρόοδος και ότι όλα έχουν ξεκαθαριστεί Εάν η πολιτική βούληση υπάρχει, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει και η χρηματοδότηση. Πού βρισκόμαστε, μπορείτε να πείτε νούμερα αναχώρα στον τομέα αυτό. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ενέργειος χώρος θεωρώ, εάν υπάρχει η θέληση, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες. Τεχνικά έχουμε τις δυνατότητες που απαιτούνται. Σημειώνω με λύπη μου ότι διάφορες ποικίλε χώρες μέλη δεν είναι, δυνατε, δεν διατεθειμένες να θεωρήσουν τόσο σημαντικά τα πλεονεκτήματα ώστε να εγκαταλείψουν κάποιες παλαιές συνήθειες. Η στρατιωτική πτυχή είναι μια πρόσθετη πτυχή το στρατιωτικό σκέλος βεβαίως παίζει ρόλο στον ενέργειο χώρο. γιατί χωρίς τη συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα δεν μπορούν να προκύψουν καν τα θετικά πλεονεκτήματα που αναμένουμε. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της επιθυμίας που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να τεθούν ενδεχομένως στην διάθεση των ε, εθνικών στατιωτικών ε, αεροποριών, πολεμικών αεροποριών, κοινοτική πόρη. Και μία ερώτηση ακόμη. Σχεδιάζει η Κομισιόν να συμπεριλάβει, να εντάξει στο ΣΕΣΑΡ πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η ΕΡΠΑΣ όπως λέγονται τώρα. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ ή κυρία Γκόμες από την Σοσιαλιστική Ομάδα. Δεν χρειάζεται να με πείσετε ότι είναι σημαντικός ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ενιαίο ουρανό. Όταν στο ε, Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε την έρευνα για τις πτήσεις της CIA το 2007. Τότε είχα συνομιλήσει με την ε, Πορτογαλική Υπηρεσία Ελέγχου του Εναέριου Χώρου και διαπίστωσα ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση, μεγάλο μπέρδεμα όχι μόνο στην Πορτογαλία και σε πολλές χώρες. <clears throat> αν ήμουν εγκληματία ή λαθρέμπορος ναρκωτικών ή λαθρέμπορος όπλων από τη Λατινική Αμερική από αλλού, πολύ εύκολα θα μπορούσα να βρω ε, χρήματα, να ε, μισθώσω ένα πολιτικό ή πολεμικό αμερικανικό αεροσκάφος, να έρθω στην Ευρώπη, να προσγειωθώ και κανένας δεν θα με ρωτήσει τίποτα. Διαπίστωσα λοιπόν ε, την μεγάλη ανασφάλεια στην οποία ε, ζούμε. Ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, μερικοί που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και από το πολιτικό και από το στρατιωτικό κλάδο υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι που είναι ανίκανοι και στους δύο κλάδους. Και οι ελεκτές εναέρες κυκλοφορίες και οι υπηρεσίες εναέρες κυκλοφορίες που έχουν άμεση σύνδεση με την Eurocontrol και που έχουν και πολιτικό και στρατικό σκέλος. Είναι πολύ ε, καλοί επαγγελματίες και τα παρακολουθούν όλα κατά Αλλά το Ινστιτούτο που υποτίθεται ότι δίνει εγκρίσεις ε, για πολιτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν <clears throat> και που πιστοποιεί, δίνει τα πιστοποιητικά σε αεροδρόμια, η δουλειά του δεν είναι και πολύ καλή. Και τη στιγμή που συμβαίνει σε μία ευρωπαϊκή χώρα, σίγουρα συμβαίνει και σε άλλη. Δεν είμαστε εμεί χειρότεροι στην Ευρώπη. Πιστεύω όμω ότι στο μεταξύ η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Σίγουρα έχει σημασία και αξία ο ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και τώρα βλέπουμε τι είδου συνεργασία υπάρχει μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου. Και βλέπετε ότι ήδη έχουμε κάποιες επιπτώσεις και στο Συμβούλιο. Γι' αυτό και το Συμβούλιο άρχισε και προβληματίζεται. Ερωτώ λοιπόν το πάνελ, τι προσπάθειες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ε, εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για το θέμα αυτό σήμερα προκειμένου να γίνει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους ώστε να μην ε, υπάρχουν τόσες επιφυλάξεις και τέτοιες αντιστάσεις που βλέπουμε σήμερα. Κάτι που προϋποθέτει και ένα καταμερισμό των κονδυλίων, γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλα ποσά. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν στις τρεις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε όλοι και στις τρεις ερωτήσεις. Μπορείτε να διαλέξετε ποια ερώτηση θεωρείτε ότι απευθύνεται σε εσά ή άπτεται των αρμοδιοτήτων του δικού σας οργανισμού. Ξεκινάμε πρώτα από τον τελευταίο μας καλεσμένο, τον κύριο Λέλο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το οικονομικό σκέλος που είναι πολύ σημαντικό όπως είπα και στην αρχή, είναι εύκολο να θέτουμε εύκολες ερωτήσεις. Και η εύκολη ερώτηση είναι πώς θα στοιχήσουν όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς εύκολη είναι η ερώτηση, δύσκολη είναι η απάντηση. Αυτό προσπαθούμε πάντως να απαντήσουμε σε αυτή την εύκολη ερώτηση. Αλλά θα πρέπει για την απάντηση να λάβουμε υπόψη 27 ε, πολεμικές αεροπορίες ε, με διαφορετικά σχέδια με διαφορετικά αεροσκάφη και με διαφορετικές αντιλήψεις για την εφαρμογή. Είναι εξαιρετικά δύσκολο λοιπόν να έχουμε έναν σαφή και ακριβή υπολογισμό. Επίσης δύσκολο είναι να συγκεντρώσουμε και τις ακριβείς πληροφορίες. Μπορούμε να στηριχτούμε όμως σε κάποιες ε, εικασίες, γενικές υποθέσεις, που φυσικά μπορούν να διαψευστούν στη συνέχεια στη φάση της εγκατάστασης. Ε, και μάλιστα αυτές οι υποθέσεις στηρίχθηκαν σε ένα μικρό αριθμό κρατών, αυτές, αυτών που έχουν τις μεγαλύτερους ε, στόλους ε, αεροπορικών σκαφών και μετά κάναμε προσωμιώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε χοντρικά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κράτη-μέλη όμως πρέπει να χρηματοδοτήσουν το όλο εγχείρημα και ο συνάδελφος θα εξηγήσει καλύτερα από μένα το πώς ε, ο μηχανισμός ε, του ενιαίου ουρανού θα λειτουργήσει. Και ο προσανατολισμός του είναι το κέρδος. Και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το, πρόγραμμα, αλλά ως επένδυση και να έχουμε και μία επιστροφή, μία απόδοση αυτής της επένδυσης και να έχουμε ένα θετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Βέβαια στην περίπτωση του στρατιωτικού κλάδου αυτό δεν μπορούν να είναι θετικό το αποτέλεσμα γιατί δεν έχουμε χρήματα. Ε, οι στρατιωτικές υπηρεσίες δεν έχουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα αυτό. Οπότε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βρουν τα κονδύλια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που δυστυχώς ε, βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Γι' αυτό και είναι σημαντική η εφαρμογή. Γιατί ίσως ε, στη διάρκεια της ε, φάσης εφαρμογής θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσουμε και το στρατητικό κλάδο που δεν έχει τόσο αποδοτικό επιχειρησιακό μοντέλο να καλύψει το κενό. Αυτό είναι σημαντικό και στη φάση του σχεδιασμού, αλλά και στη φάση της ε, εγκατάστασης, ε, όταν τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να κάνουν μια αξιολόγηση της κατάστασης και μια αποτίμηση των αναγκών τους, προκειμένου να προτείνουν κάποια σχέδια και να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτά και αφήνω το λόγο και στου υπόλοιπου καλεσμένου, Θα θέλω να προσθέσουν κάτι. Ο κύριος Μποργίνη. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Στον αφορά τις οικονομικές πτυχέ. Κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου μεταφορών που χώρα τη Δευτέρα, αναφερθήκαμε στις ανεπάρκειες του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας που στοιχίζει σε σε βάση στους Ευρωπαίους πολίτες 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, αν δείτε τις επενδύσεις που κάνουν μονομένα η στρατιωτική, ο στρατιωτικό τομέα, τότε τίθεται το ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα. Αν δούμε όμω και ποια είναι η οικονομική επίπτωση από τι ανεπάρκειε και την αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε έχετε την απάντηση. Βέβαια, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι ο μη στρατιωτικό τομέα έχει ήδη μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν πλέον τεχνολογίες οι οποίες θα είναι οικονομικά αποδοτικές και τεχνολογίες που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει και ο στρατιωτικός τομέας προκειμένου να μειωθεί αυτή η πολύ μεγάλη ζημία, αυτή η απώλεια χρημάτων 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που πλήττει τον Ευρωπαίο πολίτη. Τώρα όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας, κάναμε προτάσεις για εννιά συγκεκριμένα project, τα οποία ξεκινάνε περίπου την περίοδο αυτή. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση. Θα προσπαθούσουμε να δούμε ποια είναι τα πιθανά σενάρια για την ενσωμάτωση του άρπας στο υφιστάμενο σύστημα ATM. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για το πρόγραμμα CESAR 2020, στα πλαίσια του οποίου έχουμε ενσωματώσει και μια πιο ε, περιγραφική ε, φάση για, την, ε, για το μελλοντικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να προκύψει και θέλουμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Θεωρούμε ότι ε, τα RPAS, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ενέργειας κυκλοφορίας τα επόμενα χρόνια. Τώρα όσον αφορά τον επιμερισμό των κονδυλίων και όσον αφορά τη συμβολή των θεσμικών οργάνων. Αν καταφέρετε να δείξετε στο χρήστη ότι υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο και ότι πραγματικά υπάρχει ένα όφελο από την εφαρμογή του ΣΕΖΑΡ και ότι θα οδηγήσει σε μείωση του κόστου συστήματο, τότε αυτό είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα για να καταφέρουμε να πείσουμε του χρήστε. Η ρύθμιση από μόνη τη, οι κανονισμοί από μόνη τη δεν οδηγούν πουθενά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επιδείξουμε πρώτα τα ωφέλη του συστήματος αυτού και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του και στη θετική τεχνολογία που θα προκύψει. Από επιχειρηματικής πλευράς, ας δούμε τα πράγματα, είναι αρκετά ενδεικτικά όταν σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το ΣΕΖΑΡ το 2005-2006, οι πρώτες εκτιμήσεις ε, τότε λέγανε ότι θα έπρεπε να γίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές στα συστήματα πολιτικής αεροπορίας γιατί δεν θα μπορούσαν να αποκριθούν στα επίπεδα αυτοματοποίησης τα οποία θέλαμε να πετύχουμε. Αν απευθυνθείτε πλέον αυτή τη στιγμή στους ε, ανθρώπους που ε, αναπτύσσουν τα νέα αυτά συστήματα θα σας πούνε ότι ε, δεν χρειάζεται πλέον να τροποποιήσουν το hardware, τον εξοπλισμό, αλλά το software, τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Πάντως, η τεχνολογία Σέζαρ δεν εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο και ούτε πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα αεροσκάφη. Πάντω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αποφεληθούμε από αυτές τις τεχνολογίε προκειμένου να μειώσουμε και αυτή την απώλεια των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ξεκινήσω με το κόστος, στο οικονομικό θέμα. Δεν έχουμε καμία μαγική απάντηση για το κόστος αναβάθμισης των προδιαγραφών του ΣΕΣΕΡ. Πάντως, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι σήμερα, εξαιτίας του κατακαιρματισμού έχουμε μια αποτελεσματική χρήση του ενέργειου χώρου. Και κάθε χρόνο οι χρήστες πληρώνουν 14 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας και η επενδύσεις ετησίως είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει στραβά. Γιατί οι υποδομές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι πολύ ε, ακριβές σε σχέση με αυτά που προσφέρουν στους χρήστες. Δεύτερον, μίλησα για την κοινή χρήση των υποδομών. Έχουμε πολλές υποδομές ε, από, που είναι εθνικές, τις χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη πολεμικές αεροπορίες και υπάρχει δυνατότητα χάρη τη διαλειτουργικότητας ε, ανταλλαγής των πληροφοριών και ανταλλαγής ε, στοιχείων από ραντάρ. Βέβαια ε, αυτό προϋποθέτει μια ριζική απόφαση να δεχτεί κανείς να δώσει πληροφορίες στο, στη γείτονα χώρα ή να ε, γίνεται κοινή χρήση συστημάτων πλοήγησης. Είναι δυνατόν όμως να αναβαθμιστούμε αν πραγματικά θέλουμε και υπάρχει πολιτική βούληση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ουρανού. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε σαν για καλά εξοπλισμό εχμής ή προηγμένης τεχνολογίας ή να αντικαθιστούμε εξοπλισμό από τη στιγμή που και ο παλιός λειτουργεί ακόμη. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες υποδομές, ε, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, ιδιαίτερα για το στρατιωτικό θέμα. Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινή επιχείρηση του ΣΕΣΑΡ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και υπάρχουν ήδη, ε, υπάρχει ήδη εξοπλισμός ε, και στα αεροσκάφη και θέλουμε να δούμε τι, τι αλλαγές χρειάζονται. Οι μελέτες που έχουμε κάνει δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και μεγάλο τμήμα του εξοπλισμού των πολεμικών αεροσκαφών με μία αλλαγή του software μπορούμε να κάνουμε τις σωστές αλλαγές και προσαρμογές. Οπότε σε ό,τι αφορά την ε, συμβατότητα με τα νέα συστήματα δεν χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε όλα μας τα αεροσκάφη. Γι' αυτό μπορεί να γίνει σε μια μεταβατική περίοδο, 5-10 χρόνων. Οπότε με συνεργασία και με ενιαίο σύστημα σίγουρα θα μειώσουμε και την κατανάλωση των καυσίμων. Και τα καύσιμα είναι πολύ δαπανηρά για όλους, όχι μόνο για τις ε, αεροπορικές εταιρείες, αλλά και για την πολεμική αεροπορία. Οπότε αυτή την άποψη οι οικονομίες θα είναι μεγάλες. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες. Ενώ σήμερα μερικές φορές ε, ε, ξοδεύουμε κονδύλια και που δεν χρειάζεται. Τώρα σε ό,τι αφορά τα συστήματα μη επανδρομένων πτήσεων ή τηλεκαταστηνόμενα συστήματα αεροσκαφών. Έχουμε μόνο 14 ε, χώρες στη Eurocontrol που αποφάσισαν να υιοθετήσουν εθνική νομοθεσία για να διευκολύνουν αυτή την ένταξη των VAS. Αυτό είναι λάθος, γιατί θα έχουμε 14 διαφορετικές προδιαγραφές και 14 διαφορετικούς κανόνες, ενώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ γρήγορα να υιοθετήσει ενίους κανόνες για να επιτρέψει την ένταξή τους. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα το θέμα ε, πιστοποίησης εξοπλισμού διαχείριση ενέργειας ε, κυκλοφορίας και κοινή χρήση ε, της εμπειρογνωμοσύνης οι εποπτικές αρχές και εξειδημένες διοικήσεις θα αξιοποιήσουν καλύτερα τις υποδομές τους αν κάνουν συνεκμετάλλευση των πόρων με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό θα οδηγήσει και σε μεγάλες οικονομίες αλλά και σε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση και σύγκληση του δικτύου. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much. And last but not least, Mr. Castelletti, please. Εσείς κύριε Καστελέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική του ενιαίου ευρωπαϊκού όρανου είναι μια πρωτοβουλία που αυτό που κάνουμε με στην πολιτική αυτή είναι να αυξήσουμε την απόδοση του συστήματος, να αυξήσουμε την χωρητικότητα του συστήματος, μειώνουμε επομένω τις καθυστερήσεις, αυξάνουμε την αποδοτικότητα, την ε, ε, ικανότητα σε πτήσεις και την ασφάλεια. Άρα, καταρχήν θα πρέπει να είμαστε ικανοί να αποδείξουμε ότι τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτή την αύξηση και σε ό,τι αφορά την αύξηση της χωρητικότητας μείωση της επίπτωσης των περιβάλλων και ούτω καθεξής θα αντισταθμίσουν το κόστος της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών καθώς και το κόστος λειτουργίας των τεχνολογιών αυτών. Στην ε, αρχή της ε, φάσης εφαρμογής όπου το ΣΕΖΑΡ είναι τμήμα του ΣΕΣ θα πρέπει να μπορεί να φανεί αυτό. Για να το πράξουμε αυτό βέβαια οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση όχι μόνο το, του ωφέλους αλλά και του κόστους. Γιατί αν δεν είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε την αξιολόγηση των ωφελών δεν θα, θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα τα οποία δεν θα είναι ισχυρά. Όταν προσπαθούμε να βάλουμε ένα κόστος στο ε, ATM Master Plan στο τέλος της διαδικασίας ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ποσοτικοποιήσουμε την επίπτωση στο στρατιωτικό τομέα. Γι' αυτό το αφήσαμε ανοιχτό. Και άρχισε μια προσπάθεια μαζί με την European Defense Agency να δούμε αυτές οι τεχνολογίες τι επίπτωση μπορεί να έχουν στο στρατιωτικό κλάδο σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων σε ποια τμήματα του στόλου έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε με ποσοτικούς όρους καθαρά το κόστος την οικονομική δηλαδή επίπτωση στο στρατιωτικό κλάδο. Και όπως σας είπαν περίπου ανέρχεται το κόστος αυτό στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως αναφέρεται σε ολόκληρο το master plan. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να επιλέξουμε ένα υποσύνολο τεχνολογιών που θα εφαρμοστούν από του χρόνου και μέχρι το 2020. Και για αυτές υπάρχει, μάλλον, υπάρχει ανάγκη να γίνει ειδική ανάλυση κόστους ωφέλους. Για την περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό κόστους ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για, που θα βαρύνει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς στην βάση τιμών του 2012. Για την πρώτη φάση λοιπόν θα είναι μικρότερη αυτή και επομένω λιγότερο δαπανηρή. Και βρισκόμαστε σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για να δούμε από αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια τι, ποιο ποσοστό θα βαρύνει τον στρατιωτικό τομέα. Όταν θα έχουμε λοιπόν ξεκάθαρη εικόνα, μπορούμε να δούμε τότε πώς θα, καλύψουμε το κόστος αυτό. Μελετούμε διάφορες δυνατότητες. Από του χρόνου θα διαθέτουμε προϋπολογισμό από την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Θα έχουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια από την ευρωπαϊκή πλευρά. Τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά για να καλύψουν τα αρνητικά τμήματα του, της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Γιατί δεν είναι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν και άλλοι χρήστες. Για παράδειγμα, η αεροπορία business μπορεί να αντιμετωπίσει τις ίδιες δυσκολίες, δηλαδή αρνητική ανάλυση κόστους-οφέλους. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα οικονομικά κίνητρα για να μετριάσουμε την αρνητική επίπτωση σε ορισμένους χρήστες. Για το Pass βρισκόμαστε στην φάση σύνταξης μιας ανακοίνωσης που μάλλον θα δημοσιευτεί τις επόμενες εβδομάδες. για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων τηλεκατευθυνόμενων μη επιδρομένων σκαφών. και αυτά σε δύο επίπεδα. Αφενός στο ρυθμιστικό επίπεδο με την έγκριση συγκεκριμένων κανόνων που θα επιτρέψουν την ένταξη αυτών των αεροσκαφών διότι βέβαια όταν μπαίνουν σε μεικτό περιβάλλον τα αεροσκάφη αυτά ασφαλώς αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια και για να γίνει με ασφάλεια χρειάζεται, χρειάζονται και διαδικασίες πιστοποίησης. Δεύτερη πτυχή για την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Θα πρέπει να παρέμβουμε και σε αυτή την έρευνα και όπως σας εξηγήθηκε νωρίτερα διεξάγονται συζητήσεις με το SJU για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από του χρόνου και στο πλαίσιο αυτό η εμπειρία του στρατιωτικού κλάδου πρέπει να ληφθεί υπόψη πλήρως διότι Αυτά τα μη επιδρομένα αεροσκάφη έχουν εξελιχθεί κυρίως για στρατιωτικά. Τώρα υπάρχουν βέβαια και παρόμοιες απαιτήσει από το μη στρατιωτικό τομέα. Μιλούμε για αεροσκάφη που θα χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς, με διαφορετικό payload επομένως. Πρέπει να βασιστούμε όμως την εμπειρία των στρατιωτικών για να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πρότυπά τους, τις διαδικασίες τους, τις απαιτήσει τους που ήδη έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία από το στρατιωτικό τομέα. Να δούμε δηλαδή αν είναι δυνατόν να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των όσων ήδη γνωρίζουν και έχουν αναπτύξει οι στρατιωτικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσετε για το σχέδιο αυτό που θα εξυγχρονίσει και θα αναδιαρθρώσει τον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο. Να είστε βέβαιοι ότι εμεί ε, θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στη διαδικασία και κατά πάσα πιθανότητα θα σα ξαναπροσκαλέσουμε και στο μέλλον για να μα δώσετε περαιτέρω πληροφορίε για την πορεία τη διαδικασία αυτή. Τρίλεπτη διακοπή, αγαπητοί συνάδελφοι, και κατόπιν ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλέου θα συνεχίσει τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το επόμενο σημείο της ημερησίας μας διάταξης είναι εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης και σχετικών τροπολογιών για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική του διαστήματος. Η Επιτροπή είναι η αρμόδια επί της ουσίας για τον φάκελο αυτό. Το αρχικό έγγραφο είναι μια ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013. Ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα είναι ένας νέος τομέας στην συνθήκη της Λισαβόνας. Από γεωστρατηγική άποψη, η ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα έχει μεγάλη σημασία, διότι επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ανεξάρτητα μέσω της ανάπτυξης μιας αυτόνομης ικανότητας για δράση στο διάστημα που εμπίπτει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας να επιτύχει στρατηγική αυτονομία. Επιπλέον, οι πρόσφατες πολιτικές και στρατιωτικές επεμβάσεις ανέδειξαν τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Υπάρχουν 20 τροπολογίες συνολικά, εκ των οποίων οι 7 είναι από την εισηγήτρια. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στην, την επόμενη Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή Εξωτερικών. κυρία Κρόμπερ, έχετε τον λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δεν πρόκειται να διαβάσω τη γνωμοδότηση για τις προτάσεις, γιατί το ξανασυζητήσαμε. Θα αναφερθώ στις συμβεστικές τροπολογίες, που τελικά συμβίλησαν τις 20 ε, τροπολογίες, είναι 5 με 7. Η πρώτη τροπολογία τονίζει την στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία του διαστήματος, την ανάγκη ενίσχυση της ε, συνεργασίας και ανάπτυξη της βιομηχανικής ε, του, της βιομηχανίας του διαστήματος ε, σε συνδυασμό με, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία. Τώρα, δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα του προϋπολογισμού. Θα πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε το επίπεδο φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς και πολιτικούς μας στόχους ε, πριν συμφωνήσουμε για τα κονδύλια και εδώ στη συμβαστική τροπολογία τονίζουμε ότι η πολιτική του διαστήματος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, μεγάλο πλονέκτημα για τη συνέργεια πολιτικού στρατηγικού κλάδου αλλά και για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η τρίτη τροπολογία τονίζει ότι η συνεργασία για θέματα διαστήματος θα πρέπει να ενταχθεί στον, στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Η τέταρτη τροπολογία μιλά για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 60% των ηλεκτρονικών συστημάτων στους δορυφόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ε, τεχνολογία που εισάγουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε και τον ευρωπαϊκό τομέα γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Επίσης θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Η πέμπτη τροπολογία μιλάει για τους ε, ελέγχους εξαγωγών ε, προϊόντων διπλής χρήσης και την ανάγκη συστήματος ελέγχου και μια άλλη τροπολογία μιλάει για τα θράψματα στο διάστημα και τα διάφορα υπολείμματα που βρίσκονται σε τροχιά και ε, την αυξανόμενη χρήση του διαστήματος για στρατηγικούς λόγους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διεθνή πρωτοβουλία που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα που την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τονισμό των δραστηριοτήτων, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Και τέλος, υπάρχει ανάγκη για συνεργασία με τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για να ενισχυθεί η ειρηνική συνεργασία στο διάστημα. Αυτές είναι οι συμβαστικές τροπολογίες. Οι πράσινοι τονίσαμε το θέμα του επίπεδου των φιλοδοξιών που θα πρέπει να προσδιοριστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρούμε την ισορροπία δηλαδή, γιατί ε, αυτό το εγχείρημα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ δαπανηρό. Αλλά θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα τι εστί ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Επίσης ε, η βελτίωση της γνώσης ε, για βοήθεια αναπτυξιακή και ανθρωπιστική το θέμα του Γαλιλαίου που θα χρησιμοποιείται και για πολιτικές και για στρατιωτικές χρήσεις. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καλύπτονται από τις συμβαστικές μου τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κρόμπερ και το λόγο να έχει ο συνάδελφο Ζοχάουεν. Um, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω η τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ήταν ε, πριν την ε, προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τις τροπολογίες αυτές και να πω βέβαια στην συνάδελφό μας, την κυρία Κρόνμπερκ, ότι έχει κάνει μια πολύ καλή γνωμοδότηση, ιδιαίτερα περιεκτική και μας δόθηκε δυνατότητα χθες μαζί της να διαπραγματευτούμε με ένα πολύ ήρεμο και επικοδημητικό τρόπο τις τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της Επιτροπής μας να πούμε ότι ο στρατιωτικός κλάδος, ο στρα... η στρατιωτική συνιστόσα θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της διαστημικής πολιτικής και της βιομηχανικής διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας που έχει τόσο στρατιωτικό όσο και μη στρατιωτικό ρόλο. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με τη διαστημική πολιτική. Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες αναφερόμαστε μέσω των τροπολογιών μας στα σημεία αυτά και λέμε ότι θα πρέπει καταρχάς να αναφερθούμε πρώτα στον εξοπλισμό διπλής χρήσης. Θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται και τα προϊόντα αυτά και ξέρετε ότι θα υπάρχει σύντομα μέχρι τα τέλη του έτους μια ξεχωριστή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προϊόντα διτής χρήσης. Θέλουμε επίσης να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς όσον αφορά την διαστημική βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε να στείλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι ώστε να πλησιώνονται ρυθμιστικά σωστά όλες οι διαστημικές δραστηριότητες. Και τέλος να πούμε ότι καθώς σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα στρατηγικό πλαίσιο, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, το πλαίσιο αυτό και να λειτουργούν συλλογικά. Στις ε, χθεσινές ε, διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό ξεκάθαρα, είδαμε κάποιες τροπολογίες και είπαμε ότι θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την συνεργασία την οποία προβλέπει και η συγγήτρια. Πάντως εξ ονόματος των Βρετανών εργατικών απλώς επιβεβαιώνω αυτή τη στιγμή ότι θα έχει η συγγήτρια την υποστήριξή μας. Δεν το είπα αυτό ξεκάθαρα όταν συναντηθήκαμε χθε. Υπάρχουν κάποια διοργανικά ζητήματα. Όπως είπε και η κυρία Κρόνμπερκ υπάρχει μία απόσταση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους, αλλά αυτή θα πρέπει να καταστεί πιο στενή στο μέλλον. Θέλουμε επίσης οι οικονομικές ε, επιπτώσεις ε, να οδηγούν πραγματικά στο 7,5% οικονομική ανάπτυξη και να καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε όλα τα αδύναμα σημεία τα οποία έχει αντιμετωπίσει, τα οποία στην έκθεσή της έχει εντάξει και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Στην παράγραφο 5β αναφερόμαστε στα στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα 2020, με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, ότι θα πρέπει να προβλέπεται η απαραίτητη κοινοτική χρηματοδότηση και ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε επίση και στην αλεξάρτηση που υπάρχει με άλλε πολιτικέ και ιδίω με την πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ. Και να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και στην πολιτική αυτή και την απαραίτητη συμμετοχή τη διαστημική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη της Επιτροπής μας και είμαστε στη διάθεση της κυρίας Κρόνμπερκ, η οποία έχει καταβάλει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να συγκεράσει τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάλερ έχει τον λόγο. Yeah. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Κρόνμπερκ για την συνεργασία. Το θέμα είναι όντως τόσο σημαντικό που δεν σηκώνει ε, βαθιές διαφωνίες. Η πρόθεση των θεμάτων είναι σημαντική και για λογαριασμό της οικονομίας μας αλλά και για να ωφεληθούν όλοι οι τομείς. Συμφωνώ με τις πέντε συμβαστικές προτάσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει και όσα δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές προτάσεις εμείς υποστηρίζουμε και τις τροπολογίες 8, 9 και 10 των πρασίνων της κυρίας Κρόνμπεργκ καθώς και την τροπολογία 17 του κυρίου Χάουιτ ώστε νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε ευρεία συνένεση για τη γνωμοδότηση. Εάν θέλετε κάτι να παρέμβετε, αν θέλετε κάτι σχόλιο. Στις 24 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη, στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων θα έχουμε την ψηφοφορία. Προχωρούμε στο επόμενο μας θέμα τον Οκτώβριο του 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις που να καθιστούν σαφείς κοινέ επιχειρησιακές διαδικασίες και σαφείς κανόνες εμπλοκής για κοινέ επιχειρήσεις στην θάλασσα με στόχο την διασφάλιση της προστασίας όσων έχουν ανάγκη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2010 κάθετος 252 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στόχευσε στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, εποπτείας των θαλασσίων συνόρων, υπό τον συντονισμό του οργανισμού που συστήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η εποπτεία των θαλασσίων συνόρων κρίθηκε αναγκαία και πρόσφορη για τις μη εγκεκριμένες διελεύσεις των συνόρων, για να εμποδίζει την διασυνοριακή εγκληματικότητα και να συλλαμβάνει ή να παίρνει άλλα μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς. Οι προτινόμενοι κανόνε αυτοί καθ' αυτήν υπερβαίνουν την απλή εποπτεία και μεριμνούν για μέτρα όπω την επίσχεση πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω μέτρα είναι αναγκαία εν ώψη των συμβάντων όπου μετανάστε προσπαθούν να περάσουν παράνομα τα θαλάσσια σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαίνοντα σε μη αξιόπλοα σκάφη και συνεπώ μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση κινδύνου όταν εντοπίζονται. Άλλο στοιχείο που δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ ερμηνείε των ισχυουσών διατάξεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του διεθνού δικαίου τη θάλασσα, με αποτέλεσμα ότι σε παρόμοιε θαλάσσιε επιχειρήσει μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικοί ή ακόμη και συγκρουόμενοι κανόνε, εξού και η ανάγκη οι επιχειρήσει να συντονίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση από τον οργανισμό. Η αρμόδια για την ουσία Επιτροπή είναι λύπη με συγγητή τον κύριο Κάρλος Κουέου. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Νικολάη. Thank you, I to you. Ευχαριστώ, θα ακολουθήσω το παράδειγμά σας και θα μιλήσω κι εγώ τη δική μου γλώσσα, δηλαδή τα ρουμανικά. Έτσι λοιπόν, όπως εξήγησατε και εσείς, το θέμα είναι αρμοδιότητας της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Δηλαδή νομοθετικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την συνεργασία μεταξύ Frontex και χωρών μελών και ξεκάθαροι κανόνες για την εποπτεία, έλεγχο και κατάσχεση πλοίων σε περίπτωση παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι η απόφαση που λήφθηκε να ζητηθεί δηλαδή σχέδιο γνωμοδοτήσεως από τη δική μας Επιτροπή, η απόφαση αυτή λοιπόν λέγω ήταν ορθή. Διότι δεν μιλούμε μόνο για δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, αλλά και γενικότερα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η γνωμοδότηση βέβαια, η μορφή της γνωμοδότησης δεν μας δίνει ε, πολλές δυνατότητες γιατί είναι περιορισμένος και ο αριθμός λέξεων που έχουμε στη διάθεσή μας αλλά εγώ έχω ρίξει το βάρος μου ιδίως στην ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσω των τροπολογιών προσπαθώ να καταδείξω ότι η προστασία των θαλασσίων συνόρων είναι ουσιώδης, ιδίως για τα νευραλγικά σημεία. Επιμένω στην ανάγκη μεγαλύτερης και καλύτερης επικοινωνίας στο θεσμικό επίπεδο. Μιλώ επίσης για την ανταλλαγή πληροφοριών που θα πρέπει να διεξάγεται μεταξύ Frontex και του πυρήνα αναλύσεως των πληροφοριών αυτών που θα δημιουργηθεί. Κάνω μια προσπάθεια επίσης αξιολογήσεως των περιπτώσεων εκείνων όπου ο χώρος Σέγγεν θα επεκταθεί για να περιλάβει τη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Δύο χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Frontex και που διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα επιτήρησης των συνόρων, ωστόσο ακόμη δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν πλήρως στον Frontex. Όταν οι χώρες αυτές θα ενταχθούν στον χώρο Σέγγεν, θα χρειαστεί τότε να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Εγώ προσπαθώ τώρα να το αποφύγω αυτό. Όταν μιλούμε για ροές μετανάστευσης, συχνά μιλούν πολύ για τον χώρο της Μεσογείου. Λυσμονούν τον χώρο του εύξηνου πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, που εύκολα, μάλλον που ε, ε, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι και εκεί καταφθάνουν πολυάριθμοι παράνομοι μετανάστες. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στην επιτήρηση και προστασία του θαλάσσιου χώρου του εύξηνου πόντου. Τίθε θέμα επίσης για την κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών που παρέχουν βοήθεια σε ναυαγούς και άλλους ας είναι και παράνομοι μετανάστες. Αυτοί οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προστατευθούν απέναντι στον νόμο. Δυστυχώς, το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή είναι πολύ περιορισμένο. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι μοναχά η 19η Ενάτου. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη των εισηγητών, αλλά η διαδικασία τέλος πάντων αυτή είναι και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα ήθελα ωστόσο να σας επισημάνω ένα σφάλμα στην ε, τροπολογία υπαρθμών 9. Εκεί μιλούν για έρευνα. Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσεκ, ο οποίος δέχθηκε να συναντηθούμε χθες και χάρη στην ε, θετική συνεργασία μαζί του εξετάσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες και αντιπροσωπευτικές για την θέση της ε, υποεπιτροπής μας τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος, κύριος Λύση. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ. Μια και όλοι μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα, θα μιλήσω και εγώ πολωνικά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη, που όπως πάντα είναι πολύ πρόθυμη και συνεργάσιμη και ανοιχτή σε όλες τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις. Και, από τη στιγμή που μιλήσαμε για τον Εύξενο Πόντο, γιατί να μην μιλήσουμε και για τη Βαλτική θάλασσα. Και αυτή είναι η εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα έχουμε την Ρωσική Ομοσπονδία που δεν, είναι στην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε ροή μεταναστών από τη Λευκορωσία ή άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτή την ε, βόρεια διάσταση της Βαλτικής θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Για το θέμα της ε, προστασίας των συνόρων ε, αφορά κυρίως την ε, μετανάστευση όπως λέει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αλλά υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας ε, και εμείς ως επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το θέμα αυτό η πιθανότητα θρεμπορίου όπλων ή εμπορίου όπλων μαζικής καταστροφής ε, και διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και είναι πολλές συνεχόμενες εδώ υπηρεσίες, αλλά στην ε, προστασία των ε, συνόρων δεν έχουμε μόνο τη Frontex και τις πολιτικές υπηρεσίες, αλλά πολλές φορές έχουμε και το πολεμικό ναυτικό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία των συνόρων. Συμφωνώ με την κυρία Νικολάη ότι η υποεπιτροπή μας ε, θα πρέπει σίγουρα να συμμετέχει στην διαμόρφωση αυτού του εγγράφου χωρίς πρόβλημα θα καταλήξουμε στη συμφωνία και θα διασκεδαστούν οι περισσότερες ανησυχίες μας γιατί πραγματικά η έκθεση είναι, η γνωμοδότηση είναι πολύ καλή Ίσως ε, έμεινε μια λεπτομέρεια κάποια κρεμότητα που θα απαιτήσει περαιτέρω συζητήσεις αφορά την έκτη τροπολογία, την τροπολογία 6 και κυρίως τη διατύπωση place of safety τόπος ασφάλειας. Ίσως ε, θα πρέπει να έχουμε με ένα πιο διασταλτικό, μια πιο διασταλτικό ορισμό για το place of safety, ειδικά για κάποιους ε, που έχουν διασωθεί, γιατί θα μπορούσε να είναι το place of safety, ε, of safety σε μια τρίτη χώρα, αλλά ή σε μέρος που δραστηριοποιούνται συγκεκριμένες μονάδες. Η τροπολογία 6 λοιπόν ε, ίσως ε, χαρίζει κάποιες βελτίωσεις. Ένα άλλο θέμα αφορά την τροπολογία 9 εκεί. Προτείνουμε τη διαγραφή δύο λέξεων, το in term. Κατά τη γνώμη μου, ίσως ε, η συμπερίληψη των όρων in term δημιουργήσει παρερμηνία ή δοσυλλαβή για παρεξηγήσεις. Θα θέλαμε ε, ο κανονισμός αυτός να είναι ακριβής και γι' αυτό προτείνω διαγραφή των όρων in term στην τροπολογία 9. Έτσι θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένη διατύπωση και συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρκεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, έλθω στην ουσία, φαίνεται πως έχει γίνει ξεχωριστή διαβούλευση, αν και θυμούμε ότι είχε ακυρωθεί η συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Το Λαϊκό Κόμμα συναντήθηκε ωστόσο με άλλη πολιτική ομάδα και εγώ δεν προσκλήθηκα. Είμαι νέα στην υποεπιτροπή, ωστόσο την επόμενη φορά δηλώνει ενδιαφέρον να συμμετάσχω. Τώρα, για την ουσία. Πώς τα βλέπω τα πράγματα. Ο κανονισμός βασίζεται στα όσα έγιναν την άνοιξη του 2011 στην διάρκεια της επιβολής απαγόρησης πτήσεων στον χώρο της Λιβύης και στα χωρικά ύδατα της χώρας αυτής. Υπήρχαν όμως δεκάδες ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν επί δύο εβδομάδες να φτάσουν στην Ευρώπη και για τις δύο αυτές εβδομάδες ελικόπτερα πετούσαν από πάνω τους για να τους παράσχουν τροφή και νερό. Παρόλο που είχε επιβληθεί από τον ΝΑΤΟ απαγόρευση υπερπτήσεων, 15 άτομα τελικά έχασαν τη ζωή τους, άρα είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Φαίνεται πως δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ευθύνε μας στη Μεσόγειο. Αυτό που βρίσκω πολύ κρίσιμο εν προκειμένου είναι ότι δεν, δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκτός αυτό, δηλαδή να το αγνοήσουμε αυτό. Εάν ένα σκάφος φεύγει από τα χωρικά έδρα της Μάλτας και περνά στα χωρικά έδρα της Ιταλίας, είναι σαφές ότι πρέπει να παρακολουθείτε από τα κεντρικά της Ρώμης. Τέλος πάντων, έχουμε την... Ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μόλις αύριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή, η Υποεπιτροπή μας δηλαδή, το έθεσε το θέμα αυτό στην ημέρηση διάταξη. δεν νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα της υποεπιτροπής μας εν τέλει. Το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Frontex. Δεν έχει σχέση με εμπορικά σκάφη ή με ψαράδες. Εάν όταν μάλλον κάποιος διασώζει κάποιο πρόσωπο δεν μπορεί να κατηγορηθεί για δουλεμπόριο, διότι τέτοια πράγματα συνέβησαν στην Ιταλία. Δυστυχώς όμως δεν μιλάει εδώ κανείς για αλληλευτικά σκάφη ή εμπορικά. Επίσης, οι στρατιωτικές δυνάμεις παρέμβασης οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες. Οι κανόνες που ισχύουν για όλους δεν μπορούν να στέλνουν ανθρώπους που διασώζουν πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν δικαίωμα να τους χορηγηθεί άσυλο. Πάντως συνολικά δεχόμαστε την πρόταση γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ξανά ότι σκάφος που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης στην θάλασσα δεν μπορεί να αφαιθεί στην μοίρα του. Δεν μπορεί να βγει κανένα και να πει «Α, δεν τους θέλω άλλους αυτούς τους μετανάστες, τους αφήνω να πνιγούν». Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος, ο κύριος Πάσκου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ την μητρική μου γλώσσα, τα ρουμανικά. Φορέστε λοιπόν, παρακαλώ πολύ, τα ακουστικά σας. Όπως είπε και η ίδια η συντάκτρια της ε, γνωμοδότησης, Θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι κάπως περίεργη. Θα έπρεπε να είχε συμφωνήσει μαζί μας η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την γνωμοδότηση αυτή και από ό,τι φαίνεται τελικά σε δύο εβδομάδες μόνο θα γίνει μια συνεδρίαση. Ουσιαστικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι μια περίεργη κατάσταση. Αν αποδεχθούμε λοιπόν την κατάσταση αυτή, χωρίς να κάνουμε κάποιες επικρίσεις ή κάποιες παρατηρήσεις, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα τυποποιηθεί αυτή η κατάσταση και ανάλογες καταστάσεις θα δούμε και στο μέλλον. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα αφενός στους α, κανόνες που ισχύουν στη θάλασσα, αλλά και πέρα από τους κανόνες αυτούς, το πιο σημαντικό για μας είναι η ανθρώπινη ζωή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποια τραγικά παραδείγματα που είχαμε και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Για παράδειγμα στην Αυστραλία είδαμε κάποιες περιπτώσεις όπου καταλήξαμε σε πραγματικές ανθρώπινες τραγωδίες ακριβώς επειδή θεώρησαν οι αρμόδιες αρχές εκεί ότι οι κανόνες ήταν πιο σημαντικοί από τις ανθρώπινες ζωές. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες. νομίζω ότι θα πρέπει να συνταχθούν κατάλληλες τροπολογίες προκειμένου να επωφεληθούν όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το κείμενο. Κάθε φορά που συντάσσουμε ένα τέτοιο καονισμό επικεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο στην Μεσόγειο, γιατί άλλωστε από τη λεκάνη της Μεσογείου περνάνε τα περισσότερα μετασταυτικά ρεύματα στο δρόμο τους προς την Ευρώπη και οι περισσότερες περιπτώσεις παράνομης μετανάστευσης εντοπίζονται εκεί. Όπως, είπε και η κυρία Νικολάη, όπως το είπαν άλλωστε και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλες σημαντικές θάλασσες, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε, εκ των οποίων η κάθε μία έχει τις ιδιαιτερότητές της. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό αυτό όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών θαλασσίων περιοχών της Ευρώπης. Και ένα τελευταίο τώρα ζήτημα. Ακούσαμε ότι ε, η Ρουμανία έχει αρμοδιότητες ελέγχου χωρίς να συμμετέχει στο χώρο Σέγγεν. Πρέπει να σας πω ότι εμείς επιτελούμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και όλα αυτά τα καθήκοντα χωρίς να καταφέρνουμε να αποφεληθούμε από το, στίχη, από το σύστημα αυτό και αυτό ενδεχομένω να ικανοποιεί ορισμένου. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Με τη σειρά μου να καταθέσω κάποιες θέσεις, σύντομα σχόλια. Το πρόβλημα της παραβίασης των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σοβαρό όχι μόνο για την παράνομη διέλευση ατόμων, αλλά και για την διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωπίνων οργάνων, όπλων και οπλισμών. Η πρόταση κανονισμού είναι ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη τις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Η γνωμοδότηση της κυρίας Νικολάη ενισχύει σε γενικές γραμμές το σύστημα υποπτίας. Ωστόσο, η γνωμοδότηση παραλείπει εκτιμώ να τονίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες στο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα τις καθημερινές αφήξεις παράνομων μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία. Επίσης ιδιαίτερα επαχθείς συνθήκες για τους πληθυσμούς χωρών όπως η Συρία, ο Λίβανος και γενικά χώρες αυτές της νότιας γειτονίας που δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα για, τις, για, τα, για τα κοντινά κράτη-μέλη όπως είναι η Κύπρος, η Μάλτα, η Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν υλικά και οργανωτικά αυτά τα κράτη-μέλη, περισσότερον εποπτικά σκάφη, καλύτερα οργανωμένες υπηρεσίες στη στεριά, περισσότερα και καλύτερα μέσα και μεγαλύτερη συνοχή στην ανταλλαγή έγκαιρων πληροφοριών, σχετικά με την κίνηση υπόπτων σκαφόκοντα στην περιοχή τους. Δεν ξέρω αν κυρία Νικολάη θέλει να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ. Thank you, President. Thank you, colleague. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις απόψεις τους. Σας διαβεβαιώ ότι θα ληφθούν υπόψη περισσότερες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα στοιχεία. Καταρχήν, η δυναμική βάση αυτής της ε, γνωμοδότησης είναι η νομολογία του ΔΕΚ που είπε ότι είναι αρμόδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, θέσπιση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Το έγγραφο δεν είναι πολιτικό. Είναι τεχνικό. Γιατί το πλαίσιο αυτού του κανονισμού είναι οι κανονισμοί συνεργασίες ό,τι αφορά την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και της υπηρεσίας Frontex. Σας διαβεβαιώ ότι πολλές από τις παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη και στις διαπραγματεύσεις και την επόμενη εβδομάδα θα οργανώσω συνεδρίες των σκιωδών εισηγητών για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ προτάσεις. Λυπάμαι για την απόφαση που ελήφθη, αλλά δυστυχώ ως υποεπιτροπή της ΑΦΕΤ οφείλουμε να τηρήσουμε ε, τις ε, εντολές και δεν ξέρω τι έγινε στη συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Πάντω σα ε, διαβεβαιώ ότι θα είμαι πρόθυμη και συνεργάσιμη και με τον Γενικό Εισηγητή, τον Κατουσία Εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο και μάλιστα στη συνεδρίαση που θα οργανώσω για του σκιώδει εισηγητές θα προσκαλέσω και τον κύριο Κοέλιο για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και μαζί του και να προωθήσουμε τις δικές μας τροπολογίε. Ε, ελπίζω ότι θα περιληφθούν στη τελική έκθεση του κ. Κοέλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Νικολάη και να υπερθυμίσω ότι στις 10 Οκτώβρη θα έχουμε ψηφοφορία. Εάν η Επιτροπή επιθυμεί να παρεύει, έχει τον λόγο. Uh, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω την κυρία Νικολά για το σχέδιο γνωμοδότησης. Κάποια πολύ σύντομα σχόλια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο για επιχειρήσεις στη θάλασσα, οι οποίες θα πρέπει να συντονισμένες από την υπηρεσία Frontex, μεταξύ δηλαδή των κρατών μελών. Η πρόταση αναφέρεται στο πώς θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις αυτές, ενώ στον κανονισμό Frontex βλέπουμε πώς μπορούν να διαρθρωθούν οι επιχειρήσεις αυτές, σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να λάβουν χώρα, πού ακριβώς μπορούν να λάβουν χώρα. Όλα αυτά προβλέπονται και στο πρόγραμμα εργασίας της Frontex. Λαμβάνοντα υπόψη το ότι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτό έχει να κάνει μόνο με τι θαλάσσιε επιχειρήσει τη Frontex, οτιδήποτε έχει να κάνει με εμπορικά σκάφη βρίσκεται εκτό πεδίου εφαρμογή τη πρόταση. Και να σας πω επίσης ότι κράτη-μέλη όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κύπρος ήδη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Frontex. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης που συνέταξε η κυρία Γκόμες. Uh, Okay, περιμένουμε. Περιμένουμε λίγο. Νομίζω ότι ένα-δύο λεπτά θα είναι εδώ η κυρία. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει έρχεται σε ένα-δύο λεπτά η κυρία Γκόμες. Κέλαμ είναι εδώ. Νικολάη μόλις έφυγε. Νικολάη. Τάρατ. Δεν είναι εδώ. Να είναι η κυρία Ναι, ναι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι κάνετε στη καλά. Καλά ήταν. Πώς πέρασε το καλοκαίρι. Καλά. She's come okay. Να καλωσορίσουμε την κυρία Γκόμες. Το επόμενο σημείο λοιπόν στη ημερησία διάταξη είναι εξέταση του σχεδίου γνωμονότησης που συνέταξε η κυρία Γκόμες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Η επικεφαλής επιτροπή για αυτό το φάκελο είναι η το αρχικό έγγραφο για την ελόγω γνωμοδότηση είναι η πρόταση της Επιτροπής για την Οδηγία σχετικά με τα μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας, δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Καθώς τα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δικτύων πληθαίνουν, η ανάγκη βελτίωση της ασφάλειας του διαδικτύου, των ιδιωτικών δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Και αυτό γιατί η ασφάλεια των δικτύων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ένα αξιόπιστο περιβάλλον στον τομέα των υπηρεσιών και της οικονομίας γενικά. Σήμερα θα συζητήσουμε την προτινόμενη γνωμοδότηση με την εισηγήτρια μας, κυρία Γκόμες, η οποία επικεντρώθηκε στις κύριες πτυχές της ασφάλειας από τη σκοπιά της ΣΕΝΤΕ. Το λόγο, κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, πρόκειται για την οδηγία, για μέτρα, για την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου ασφάλειας των δικτυών σε όλη την Ένωση. Και όπως είπατε, η ΙΜΚΟ είναι η α, κυρίως αρμόδια επιτροπή. Εμείς γνωμοδοτούμε. Καλό είναι που γνωμοδοτούμε, διότι είναι σωστό να λυθεί υπόψη η δουλειά της υποεπιτροπής στη βάση του σχεδίου του συναδέλφου μας του Νεκέλαμ για την ασφάλεια των δικτύων. Εγώ ρίξα μια ματιά, κοίταξα δηλαδή, σοβαρά την ε, βασική έκθεση και θεώρησα ότι όντως πρέπει να συμμετάσχει η Επιτροπή ΣΕΝΤΕ ε, Ασφάλειας και Άμυνας. Η δική μου φροντίδα είναι να βάλουμε και την διάσταση εξωτερικής ασφάλειας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η ασφάλεια των δικτύων να γίνει αποτελεσματικότερη, να προσφέρει περισσότερα στους πολίτες. Και αυτό σημαίνει ασφάλεια πληροφοριών σε κρίσιμες υποδομές όπως προβλέπεται και στην ευρύτερη στρατηγική της Ένωσης ως τμήμα του πακέτου που υπέβαλε η Κομισιόν τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Υπάρχουν και ορισμένε τροπολογίες, με, έχω καταθέσει δηλαδή με σκοπό να διευκρινίσω ορισμένα σημεία της οδηγίας και κυρίως να, να τονίσω την ανάγκη βελτίωσης του κοινού επίπεδου ασφαλείας και της εσωτερικής ε, στρατηγικής ασφάλειας και της ασφάλειας της Ένωσης, η συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων φορέων των τομέων της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας και για παράδειγμα με συμμετοχή της ΥΠΑ της εκπροσώπου και αντιπρόεδρου της Κομισιόν στην ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα διάφορα εργαλεία. Επίσης η διεθνή συνεργασία με παγκόσμιους παράγοντες με χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες, παρόμοιους κινδύνους μιας και δεν γνωρίζει με ε, η απειλή στον κυβερνοχώρο. Επίσης κάνω αναφορή και στη ρήτρα αλληλεγγύης και αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνονται και στην θήκη της Λισαβόνας που έλειπαν αυτά τα πράγματα λόγω αυτής της στενής ε, διάστασης εσωτερικής ασφάλειας. Ίσως να σημειωθούν κάποια προβλήματα στην περαιτέρω πορεία της ε, έκθεσης και στην ΙΜΚΟ και στην ΙΤΡΕ που είναι αρμόδιες επί της ουσίας. Ελπίζω ωστόσο η γνωμοδότηση της... Ε, υπάρχει και η γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ αλλά και η δική μας γνωμοδότηση πιστεύω θα συμβάλλουν να επιληθούν ορισμένα από τα προβλήματα αυτά, αν και δεν είμαι βεβαία. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί γνωρίζω ότι ο εισηγητής στην Επιτροπή ΙΜΚΟ προσπαθεί να αφαιρέσει από το σχέδιο της Κομισιόν μια αναφορά στην εμπλοκή του δημόσιου τομέα, το οποίο για μας είναι στοιχειώδες. Εν προκειμένου αναμένω την στήριξη του κ. Κέλαμ γιατί εκεί η συγκητής είναι ο κ. Σραφ από τη δική του πολιτική ομάδα. Ίσως μπορείτε να βοηθήσετε να τον πείσουμε ότι δεν είναι σωστή ιδέα να εξαιρέσει τον δημόσιο τομέα. Αυτή είναι η σημασία νομίζω της ε, συμβολής μας, με την κινητοποίηση δηλαδή των διαφόρων πολιτικών ομάδων μέσω των εισηγητών τους και κυρίως των βασικών εισηγητών. Αυτή νομίζω είναι πιο, το πιο σημαντικό στοιχείο της συμβολής μας. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες και ο κύριος Κέλαμ έχει τον λόγο. Yes, uh, thank you very much. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συνάδελφο Γκόμες για την πολύ δημιουργική και θετική της ε, συνεισφορά μέσω της γνωμοδότησης. Κρίμα, αλλά δεν είχαμε αρκετό καιρό και δεν προλάβαμε να συναντηθούμε για να αναλύσουμε την πρότασή σας. Πάντως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συμφωνώ σχεδόν με το σύνολο των προτάσεων. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στη ρήτρα αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό να την προσθέσουμε. Γιατί θα πρέπει να την ορίσουμε πρώτα. Τι σημαίνει η ρήτρα αλληλεγγύης και πώς θα εφαρμοστεί σε νέες καταστάσεις όπως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή τέτοια κυβέρνο Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεργασία και την ε, συνεκμετάλλευση, κοινή χρήση, πολύ σημαντικά. Και ε, βρήκατε δουλειά και για τις αρμόδιες υπηρεσίες ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μικροπροβλήματα τώρα για τις τροπολογίες 12 και 14. Εκεί αντικαταστήσατε ε, το ευαίσθητα και εμπιστευτικά από το διαβαθμισμένα και μη διαβαθμισμένα. Είμαι κάπως επιφυλακτικός, γιατί αν μιλούμε για διαβαθμισμένες ε, πληροφορίες, Εννοούμε απόρριτα εθνικής ασφάλειας, εθνικά μυστικά ουσιαστικά. Οπότε αν θέλουμε κοινή χρήση των πληροφοριών, δεν μπορούμε να μοιραστούμε ε, πληροφορίες ε, που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Σίγουρα όχι. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε την ορολογία που χρησιμοποιούμε εδώ. Δεύτερο πρόβλημα αφορά την τροπολογία 18 το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης. Συμφωνώ με το πρώτο τμήμα ότι θα πρέπει να έχουμε αιτήσει έκθεση για τα διάφορα σημεία περιστατικά, αλλά για το Β έχω κάποιες εμφιβολίες. Σαν να παρατραβάμε τις δυνατότητες που έχει η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε δύο εβδομάδες να κάνουν ενημέρωση αν κάτι συμβεί σε σχέση με μια τρίτη χώρα. Θα προτιμούσα το εδάφιο Β του 18 να διαγραφεί και να μείνουν το Α και το Γ. Τώρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα θα συναντηθώ με τον καθήλιο αρμόδιο συγγετή, γιατί η οδηγία αφορά τους παρόχους υπηρεσιών στην αγορά και τις κρίσιμες υποδομές. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η δημόσια διοίκηση πολύ συχνά υστερεί σε ό,τι αφορά το βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Επίσης, υπάρχει το θέμα της εμπιστοσύνης και της αμοιβαιότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να το επισημάνουμε και να φροντίσουμε ώστε οι δημόσιες διοικήσεις να εφαρμόσουν το ίδιο επίπεδο ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας για να αποφευχθούν παραβιάσεις ε, της ασφάλειας. Οπότε απαιτούμε κάτι από τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει το ίδιο να ζητούμε και από το δημόσιο τομέα. Να είναι έτοιμος και ο δημόσιος τομέας να κάνει κάτι αντίστοιχο. Γιατί μπορεί στα χαρτιά να φαίνεται αυτό εύκολο, αλλά στην ουσία έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη. Καλά. Από την Επιτροπή, υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση. Thank Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι επικεφαλής της μονάδας Trust and Security της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια και για την οδηγία AINIS. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, αλλά από την άλλη να εκφράσω και κάποιες αμφιβολίες ως προς το αν είναι σκόπιμο να ενταχθεί ο κλάδος της άμυνας και της ασφάλειας στην πρόταση. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πρόταση αυτή, η νομική βάση της πρότασης αυτής είναι το άρθρο 141 της συνθήκης, που ουσιαστικά είναι η νομική βάση για την εσωτερική αγορά. Στόχος λοιπόν της πρότασης είναι να εξασφαλίσουμε ότι το δίκτυο και τα επιμέρους συστήματα τα οποία βρίσκονται στη βάση κάποιων σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών διαδικασιών, τα οποία είναι ιδιαίτερα ουσιώδη για τη λειτουργία της ιστορικής ε, αγοράς, είναι αρκετά ανθεκτικά και ασφαλή. Η οδηγία λοιπόν, βασικός στόχος λοιπόν της οδηγίας, είναι να εξασφαλίσει την ε, συνέχεια των ε, υπηρεσιών αυτών, όπως για παράδειγμα κατανομή και φοδιασμός σε φυσικό αέριο, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ψηφιακών εξοπλισμών που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ψηφιακή ατζέντα. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μέσω της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των δικτύων και μέσω βέβαια της λειτουργίας των δημοσίων αρχών που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα. Το ζήτημα λοιπόν αυτής της απρόσκοπτης λειτουργία και της συνέχειας βρίσκεται πραγματικά στο κέντρο τη πρόταση αυτή, και ενδεχομένω να υπάρχουν και κάποιε δευτερογενέ επιπτώσει στη συνέχεια, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο σύστημα, καθώς επίσης και η αποφυγή οποιοδήποτε, οποιασδήποτε εγκληματική ενέργεια στα πλαίσια του κυβερνοχώρου. Ουδέποτε όμως, επεξεργαζόμενοι την πρόταση αυτή και βάσει της νομικής βάσης, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει το πεδίο εφαρμογή να διευρυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συμπεριλαμβάνει τον αμυντικό τομέα, το στρατικό τομέα, γιατί συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της συνθήκης ξέρετε ότι η αμυντική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα γίνει, ε, οποιαδήποτε αλλαγή δηλαδή, δεν θα γίνει αποδεκτή εύκολα από το Συμβούλιο. Ως προς αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εν λόγω οδηγία αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις αρχές του έτους και παρέχει κατά αυτόν τον τρόπο μία στρατηγική που έχει ένα μη στρατιωτικό σκέλος, το δικό μας δηλαδή σκέλος, και ένα σκέλος το οποίο έχει να κάνει με την επιβολή του νόμου και ένα σκέλος το οποίο έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια. Και εκεί πέρα αναφερόμαστε περισσότερο στην εξωτερική διάσταση της ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και για το σκέλος αυτό ασχολείται πιο άμεσα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θέλουμε ουσιαστικά να εκμεταλλευτούμε τις πιθανές συνέργειες ανάμεσα σε όλα αυτά τα σκέλη και τους παράγοντες οι οποίοι ενεργοποιούνται στα σκέλη αυτά, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Μολονότι λοιπόν ισχύει η πτυχή αυτή, δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποιο λόγο ότι είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή οδηγία για να συμπεριλάβουμε το στρατιωτικό αμυντικό τομέα. Δύο ακόμα παρατηρήσει, ε, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, η διαχείριση του κινδύνου, καθώς επίσης και η επιβολή αναφορών ως προς τα διάφορα συμβάντα στα πλαίσια της οδηγίας, έχουν να κάνουν μόνο με τους λεγόμενους market operators, τους παράγοντες δηλαδή στο πλαίσιο της αγοράς, τους ε, φορείς ε, εκμετάλλευσης που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες ιδίως ε, αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών όπως το Facebook ή Google δεν ισχύουν οι διατάξεις αυτές, δηλαδή η διαχείριση του κινδύνου και η αναφορά συμβάντων δεν έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν software ή με αυτού οι οποίοι ασχολούνται με το hardware. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, αυτό θα βάρει όλο ιδιαίτερο στι εταιρείε του. Και δεύτερον, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά είναι ευκταίο, είναι όντω επιθυμητό να γνωστοποιούμε, να κοινοποιούμε ένα σφάλμα το οποίο είναι γενές σε ένα πρόγραμμα λογισμικό ή σε έναν εξοπλισμό, σε ένα hardware. Γιατί στη συνέχεια ενδεχομένως ο κατασκευαστής να μην είναι σε θέση να διορθώσει το σφάλμα αυτό. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Πάντως αν συνέβαινε κάτι τέτοιο αυτό θα αύξανε το επίπεδο ανασφάλειας ουσιαστικά θα στιγμάτιζε αρνητικά τις εταιρείες αυτές που αναπτύσσουν το εν λόγω software ή hardware. Και μια τελευταία παρατήρηση. Η εισηγήτρια μας είπε πιο συγκεκριμένα στην τροπολογία 18, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει μια νέα έκθεση, θα παράσχει μια νέα έκθεση όσον αφορά τα συμβάντα τα οποία έχουν προκύψει, η οποία θα πάει προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνει καμία απολύτως τέτοια έκθεση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα σύστημα κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα διάφορα συμβάντα ουσιαστικά κοινοποιούνται στα κράτη-μέλη μέσω των ίδιων των εταιριών εκείνων που συμμετέχουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Εμεί δεν είμαστε αποδέκτε καμία τέτοια κοινοποίηση. Θα ήταν αδύνατο να χειριστούμε άλλωστε τέτοιε κοινοποίησει εκτό και να τροποποιήσουμε εντελώ τελικά την οδηγία. Θα ήταν αδύνατο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να χειριστεί τέτοιες, τέτοιο εντοπισμό συμβάντων και τέτοιε εκθέσει. Το πολύ και το λόγο έχει η ΕΕΣ. Uh, good afternoon. Uh, Λέγομαι Μακλάρεν και εργάζομαι στο τμήμα πολιτικής κυβερνοχώρου της ΕΕΣ. Όπως είπε ο Τζουζέπε, αναπτύξαμε τη στρατηγική μαζί σε συνεργασία με τη g και τη G-Connect ως μέρος στρατηγικής που ε, ε, επεξεργάζεται και θέματα άμυνας ως ενίο πακέτο από την αρχή αφήνοντας τα πιο εθνικά θέματα που αφήνουν οι συνθήκες στον χώρο αρμοδιότητας των χωρών μελών, αφήνοντα τα λοιπόν στις χώρες μέλη, αλλά ταυτόχρονα προωθώντας κάποιες συνέργειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη στρατηγική μας δίνουμε ένα μεγάλο μέρος στην κυβερνοάμυνα. Υπάρχει και ομάδα project κυβερνοάμυνας που απαρτίζεται από όλες τις συμμετέχουσες χώρες μέλη, από προσώπους τους δηλαδή, και στα πλαίσια αυτά οι, οι ικανότητες των χωρών μελών μπορούν να αναπτυχθούν και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις ενισχύσει με χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών κλπ. Πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα και είναι δύο διαφορετικές διαφορετικοί χώροι αρμοδιότητας γιατί το άλλο τμήμα είναι της ενιαίας αγοράς και θα πρέπει να μην χωριστεί. Όμως ...ο οδηγία NAS είναι σημαντική για την εθνική ασφάλεια των χωρών μελών διότι γνωρίζουμε ότι 80% της κρίσιμης υποδομής λειτουργείται από τον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις χώρες μέλη και εμείς αναλύουμε την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα που είναι μεγάλη σημασία για τις χώρες μέλη και ιδίως εκείνε που δεν είναι ακόμα αρκετά καλά προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν απειλές των κυβερνοχώρων. Γι' αυτό η οδηγία αποτελεί μια πολύ θετική ε, συμβολή στις ευρωπαϊκές ε, οδηγίες ε, που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την συνειδητοποίηση για τις απειλές στον κυβερνοχώρο στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε αντιλαμβάνομαι η κυρία Γκόμες θέλει να μιλήσει. I Ναι, κατανοώ και ε, κατανοώ ε, τον καταμερισμό έργου μεταξύ Κομισιόν και ΙΕΣ που έχετε θεσπίσει για τακ, λόγους τακτικής για να ξεπεράσετε τη διστακτικότητα ίσως κάποιων χωρών μελών αλλά μιλούμε για διαφορετικές πτυχές του ίδιου πράγματος που πρέπει να ενωθούν. Κάποιος πρέπει να το τονίσει αυτό. Την ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πράξει το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον η παρούσα υποεπιτροπή. Ίσως στο τέλος η πλειοψηφία να το απορρίψει. Θα δούμε. Αλλά δεν νομίζω να γίνει και καμιά ζημιά αν η υποεπιτροπή μας το προωθήσει. Αν και όπως είπα, κατανοώ ότι ίσως να μην αποδειχθεί πολύ δημοφιλές, πολύ δημοφιλής αυτή η προσπάθεια. Πιστεύω λοιπόν ότι οι απόψεις που καταθέτω εδώ, καθώς επίσης τις μοιράζεται και τον Εκέλαμ, είναι σωστές. Αν και Κατανοώ ότι μπορεί να μην γίνουμε κατανοητοί, αυτό το πω έτσι, στην φάση αυτή. Πολλά ακόμη πράγματα μπορούμε να ρυθμίσουμε. Τα προβλήματα δηλαδή που ανέφερε ο Τούνε Κέλαμ σχετικά με την διατύπωση, την ορολογία καλύτερα, διαβαθμισμένες, εμπιστευτικές, που άπτεται ακριβώς του άλλου στοιχείου που εξηγήσατε ως πρόβλημα, τους κανόνες του Κοινοβουλίου δηλαδή, μπορούμε να βρούμε και εκεί κάποια λύση μεταξύ μας, καθώς επίσης και στο θέμα της υποβολής αναφορών. Υπάρχει Βέβαια και μια ευρωπαϊκή αρχή την οποία θεσπίζει η οδηγία υπό την αιγίδα της Κομισιόν, έτσι δεν είναι. Αυτή η ευρωπαϊκή αρχή που δημιουργείται οδηγία, ποιος, ε, ποιος, ποιος την χειρίζεται αυτήν. Αυτή ήταν ε, εσκεμμένη επιλογή δεν δημιουργούμε νέο οργανισμό, νέα υπηρεσία ή αρχή, αλλά ένα δίκτυο. Δίκτυο αρμόδιων αρχών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετέχει με γραμματιακή υποστήριξη στο δίκτυο και θα καθορίσουμε τους κανόνες της διαδικασίας για τη, για τη λειτουργία του δικτύου στα κράτη-μέλη. Και επίσης επειδή στο δίκτυο τα κράτη-μέλη θα ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και θα ενημερώνονται για διάφορα συμβάντα, θα γίνεται ενημέρωση για τα συμβάντα αυτά. Όλα αυτά θα γίνουν με χρήση ασφαλούς υποδομής. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη θα καθορίσει ποιες είναι οι προδιαγραφές ή προϋποθέσεις για την ε, ε, εισαγωγή ενός κράτους σε αυτή την ασφαλή υποδομή. Αλλά δεν έχουμε νέα αρχή, δεν δημιουργείται νέα αρχή. Όπως είναι το σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστικών, Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής για τις Τηλεπικοινωνίες. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο. this... Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ο Τούνα, εγώ και άλλοι συνάδελφοι καλό θα ήταν να βολιδοσκοπήσουμε και τους υπόλοιπους για να δούμε τι γνώμη έχουν για το σημείο αυτό. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο προσεκτικοί, τόσο διστακτικοί όσο η Επιτροπή. Γιατί θέλουμε πρόοδο σε κάτι που θα διευρύνει τις ικανότητες και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο. Απ' την άλλη γνωρίζουμε ότι μόνο μια σφαιρική προσέγγιση, μια ολιστική προσέγγιση θα μπορέσουμε να εντάξουμε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και μόνο έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα και στο Κοινοβούλιο και ειδικά στην υποεπιτροπή μας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εμείς να δείξουμε το δρόμο κατά κάποιο τρόπο ακόμη και αν δεν συμφωνούν όλοι γι' αυτό. Πάντως το σημαντικό είναι μεταξύ μας τουλάχιστον οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουμε, να συνεννοηθούμε ώστε να δώσουμε μία γνωμοδότηση της υποεπιτροπής που θα είναι συνενετική στο μέτρο του δυνατού. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες. Απλά δύο υπενθυμίσεις ότι μέχρι τις 26 του Σεπτέμβρη θα έχετε δυνατότητα κατάθεση τροπολογιών και η επόμενη μας συνεδρία θα είναι 25 με 26 του Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πολύ. Έκλεισε η συνεδρία.